Euh, Καλημέρα σας. Θα ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας λοιπόν. Ε, δέχεστε τη μερισία διάταξη, έχετε να κάνετε κάποιο σχόλιο. Πήρατε τα πρακτικά της συνεδρίασης της 3ης Μαρτίου 11. Εάν έχετε παρατηρήσει σχετικά με τα πρακτικά, πρέπει να καταθέσετε τις παρατηρήσεις πριν από τις 12.30, αλλιώς θεωρούνται δεκτά. Τώρα για το λεπτό των ερωτήσεων. Πήραμε από πλευράς της κυρίας Κέλλερ και Φαγαντίνη μια ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προς την Επιτροπή μάλλον για τη συνεδρίαση αυτή. Πριν δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την απάντησή σας, ε, μετά την απάντηση της Επιτροπής μόνο αυτοί που κατέθεσαν την ερώτηση μπορεί να καταθέσουν μια συμπληρωματική σύντομη και εφόσον συνδέεται άμεσα με την αρχική συζήτηση και την απάντηση της Επιτροπής. Το λόγο λοιπόν έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Απαντώντας στην ερώτηση Κέλλερ και Σατζεντίνη. Είναι παρούσα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Euh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόκειται για τέσσερις ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και οι τέσσερις αναφέρονται στο θέμα των πρώτων υλών. Η πρώτη ερώτηση ρωτά τον τρόπο με τον οποίο η στρατηγική για τις πρώτες ύλε η οποία υιοθετήθηκε το 2008 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συμπληρώθηκε στις αρχές του 2011 μέσω μιας νέας ανακοίνωσης πώς λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα και τις ανάγκες των υποανάπτυξη χωρών. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και οι δύο ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καλύπτουν τους δύο βασικούς πυλώνες, από τη μία δηλαδή την προβληματική της πρόσβασης στις πρώτες ύλες, κάτω από ισότιμες συνθήκες, και εκεί περιλαμβάνεται αν θέλετε το βιομηχανικό κομμάτι πάνω στο οποίο έχουμε κάνει πολλές συζητήσεις. Ο δεύτερος πυλώνας όμως αφορά την προβληματική της ανάπτυξης και ιδιαίτερα τα συμφέροντα και τα προβλήματα των εταίρων μας που αντιμετωπίζουν οι εταίροι μας η υποανάπτυξη χώρες. Στο πλαίσιο αυτό η στρατηγική που ακολουθήσαμε ήδη από το 2008 προτείνει διάφορους άξονες παρέμβασης. Καταρχάς την ενίσχυση των δυνατοτήτων των υποανάπτυξη χωρών, οριζόντιος βασικός στόχος μας, κάτι το οποίο αφορά συνολικά το θέμα και το θέμα των πρώτων υλών. Δεύτερον, την δημιουργία ενός ε, επενδυτικού κλίματος ευνοϊκού με στόχο την αύξηση της διαφάνειας των συμβάσεων συμβολέων στον τομέα των εξορρυκτικών δραστηριοτήτων και ταυτόχρονα τον καθορισμό ενός δικητικού και ε, νομικού πλαισίου αποτελεσματικού, όπως επίσης και τον καθορισμό ενός πλαισίου φορολογικού σε σχέση με τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με, την, με τα μεταλλεύματα κτλ. Συνεπώς, ο τομέας αυτός αντιμετωπίζεται πάρα πολύ συχνά λοιπόν στα πλαίσια των λεγόμενων οριζόντιων πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακόμα και όταν οι τομείς αυτοί δεν ονοματίζονται θα έλεγα συγκεκριμένα. Ε, περνώ τώρα στην τέταρτη, αν μου επιτρέπετε, των τεσσάρων ερωτήσεων που αφορά τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι προφανές ότι όπως και σε όλες τις άλλες πολιτικές, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών κανόνων και του κράτους δικαίου είναι βασικές αρχές που διέπουν τη συνεργασία μας με τις υποανάπτυξη χώρες. Όχι λοιπόν γιατί επειδή ο συγκεκριμένος τομέας δεν αντιμετωπίστηκε συγκεκριμένα στα πλαίσια της πολιτικής για τις πρώτες ύλες, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν εφαρμόζονται οι γενικές αρχές που εφαρμόζονται σε όλους τους τομείς, σε όλες τις επιχειρήσεις και σε όλες τις δραστηριότητες, πόσο μάλλον και στην εξαγωγή μεταλλευμάτων και πρώτων υλών και την εκμετάλλευσή τους. Λοιπόν, δεν αφιστάμεθα συνεπώς των βασικών αρχών και των θετικών κανόνων που ήδη υπάρχουν και συνεπώς οι συμφωνίες τις οποίες έχουμε συνάψει με πολλές από τις υποανάπτυξη χώρες, οι συμφωνίες αυτές περιλαμβάνουν ρήτρες για τα ανθρώπινα δικαιώματα και με συνέπεια εφαρμόζονται και στον τομέα των πρώτων υλών. Έρχομαι τώρα προς τα πίσω στην ερώτηση παρίθμου 2 διαρωτάται η, ε, ε, η, η κυρία που κατέθεσε την ερώτηση αν η στρατηγική περιλαμβάνει επίσης πιθανές κυρώσεις σε σχέση με τις χώρες οι οποίες θέλουν να επιβάλλουν περιορισμού στην εμπορία, εξαγωγή, εισαγωγή πρώτων υλών. Και στην περίπτωση αυτή, εάν αυτό είναι συμβατό με την αποτελεσματικότητα της βοήθειας και το άρθρο 208 της, πολι... της Συνθήκης της Λισαβόνας. Η στρατηγική δεν προβλέπει καμία κύρωση. Πρόκειται για στρατηγική, ένα policy document ουσιαστικά. Δεν είναι το κατάλληλο εκτελεστικό μέσο, αν θέλετε, για την επιβολή κυρώσεων. Αυτό είναι κάτι το οποίο σχεδιάζεται σε ένα ξεχωριστό και ανεξάρτητο νομικό πλαίσιο. Γι' αυτό λοιπόν δεν υπάρχει αναφορά στις κυρώσεις. Άλλωστε θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύει ότι στις περισσότερες, σε κάποιες περιπτώσεις και ιδιαίτερα σε προσωρινό χρονικό διάστημα κάποιοι περιορισμοί θα μπορούσαν και να τεκμηριωθούν. Ε, είναι κάτι το οποίο είχε τεθεί στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων για την οικονομική εταιρική σχέση με τις χώρες ε, ΑΚΕ και πάρα πολύ συχνά εκεί είδαμε, αλλά για προσωρινό χρονικό διάστημα, και θυμίζω ότι έτσι και αλλιώ οι συμφωνίες αυτές δεν έχουν τεθεί σε λειτουργία ακόμα, αλλά μπορούμε να βρούμε κάποιες προσωρινές λύσεις που να εικονοποιούν τα συμφέροντα των χωρών που είναι συμβαλόμενες με εμάς. Παραμένοντας ευέλικτη λοιπόν στον τομέα των περιορισμών στις εισαγωγές, Παραμένει το θέμα εάν οι συγκεκριμένες μορφές περιορισμού είναι αποτελεσματικές σε σχέση με τον στόχο του σαν μέσα. Έχουμε πάρα πολλές αμφιβολίες ως προς αυτό και θεωρούμε ότι θα πρέπει να εξετάσουμε με πάρα πολύ προσοχή τις συγκεκριμένες περιπτώσεις στα πλαίσια των οποίων θα μπορούσε να δικαιολογήσει κανείς τέτοιου είδους περιορισμού στις εισαγωγές αλλά επαναλαμβάνω ότι κάποιες προσωρινές εξαιρέσεις ε, θα μπορούσαν να καλύψουν τις πραγματικές ανάγκες των υποανάπτυξη χωρών. Να προσθέσω εδώ ότι συχνά οι περιορισμοί αυτοί παίρνουν μορφές οι οποίες δεν είναι σεμβατές με τις ισχύουσες συνθήκες είτε του ΠΟΕ είτε της διμερείς συμφωνίες Οπότε σε αυτή την περίπτωση είναι αυτονόητο ότι όταν υπάρχουν παραβιάσεις συγκεκριμένων ισχυουσών συμφωνιών, τότε τίθεται το θέμα ε, σε τις θέσεις σε λειτουργία της διαδικασίας επίλυσης διαφορών. Παραμένει ένα τρίτο θέμα. αφορά την, ή μάλλον η τρίτη ερώτηση ήταν για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όχι η τέταρτη όπως σας είπα, έκανα λάθος. Περνάω τώρα στην τέταρτη. Ε, θα μείνω εδώ, θα περάσω στην αγγλική γλώσσα γιατί πρέπει να είναι κανείς επακριβής νομίζω σε αυτό το τέταρτο θέμα της ε, ε κυρίας που έθεσε τις ερωτήσεις. Στόχος μας είναι να υπάρξει ένας απορριθμισμένος ε, χώρος για την ανάπτυξη της ελεύθερης αγοράς. Σε ένα τέτοιο χώρο πόσο μπορεί η πολιτική για τις πρώτες ύλε να είναι συνεκτική με την αναπτυξιακή ε, ε, βοήθεια. Πώς είναι δυνατόν να γίνει αυτό. Υπάρχει εδώ μια παρανόηση σε σχέση με το περιεχόμενο και τον στόχο των ανακοινώσεων της Κομισιόν. Δεν νομίζω ότι λέγουμε εμείς σε καμία περίπτωση ότι στόχος μας είναι να δημιουργήσουν μια μη διακανονιζόμενη και απόλυτα φιλελευθεροποιημένη αγορά. Οπότε δεν χρειάζεται να σχολιάσω, αν θέλετε, την υπόθεση αυτή, η οποία είναι προϊόν μάλλον παρανόησης και δεν χρειάζεται εξηγήσεις. Θα ήθελα να επανέλθω ε, τους ε, κυρώσεις ή τους περιορισμούς όπως τους χαρακτηρίσατε και είπατε ότι μπορεί να είναι σε ορισμένες περιπτώσεις προσωρινές. Πότε πιστεύετε ότι είναι αιτιολογημένες και πότε όχι και ποιες, ε, ποιους περιορισμούς έχει κατά νου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν ομιλεί για κυρώσεις ή για περιορισμούς ακόμη και αν δεν αναφέρονται σε αυτό το έγγραφο έγγραφο. Πότε υπάρχουν ε, περιορισμοί ή κυρώσεις και πότε είναι αιτιολογημένες. Για δύο λεπτά μόνο λέει η Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Θα πάρω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα το οποίο έχω επεξεργαστεί. Είναι η προετοιμασία της συμφωνίας ε, για τις χώρες ΣΑΝΤΕΚ ε, του χώρου της Αυστραλίας εκεί είχαμε δεχθεί να συζητήσουμε προσωρινά, διότι ακόμη δεν έχουμε συνάψει τη συνθήκη, ε, την αρχή είτε να υπάρξει καταβολή εξαγωγικών φόρων ή ποσοστώσεων που σε μια μορφή που ακόμη δεν ε, έχει εξεταστεί και ε, αυτό όταν πρόκειται για νέες επενδύσεις οι οποίες πρέπει να προωθηθούν χωρίς όμως να υπάρχει ατέρμον διάρκεια διότι ε, μπορεί μία επένδυση να στηριχτεί για 5-10 χρόνια όχι για όλη τη διάρκεια της για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος και ε, έχουμε βέβαια και άλλα μέσα για να προστατεύσουμε το περιβάλλον, αλλά είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τα επιχειρήματα υπέρ ορισμένων ε, εξαγωγικών περιορισμών που αιτιολογούνται βάσει της προστασίας του περιβάλλοντος. Πιστεύω ότι αυτά είναι τα δύο βασικά επιχειρήματα. Είχαμε εξετάσει διάφορες ε, ε, λύσεις, αλλά εφόσον δεν υπάρχει ακόμη κύρωση ή υπογραφή συμφωνίας, δεν χρειάζεται να προχωρήσουμε περαιτέρω και οι δύο βασικές προϋποθέσεις που είχαμε εξετάσει ήταν οι νέες ε, επενδύσεις και το περιβάλλον. Ευχαριστώ. Στο θέμα τώρα ε, των ανακοινώσεων της Προέδρου θα ήθελα απλώς να αναφερθώ ε, στα πολύ ε, σοβαρά γεγονότα στην Ιαπωνία, στη Φοκουσίμα και τον κίνδυνο για τον παγκόσμιο πληθυσμό άρα αντιλαμβάνεστε πόσο σοβαρή είναι η θέση των χωρών των υποανάπτυξη, του, των υποανάπτυξη χωρών και επίσης ε, θέλω να ε, σκεφτώ και την ε, θέση ε, του, των Ιαπώνων μέσα στις, σε αυτούς τους πυρηνικούς σταθμούς υπάρχει πλουτόνιο το οποίο δεν αποσυνδέεται παρά μόνο μετά από δεκάδες εκατομμύρια χρόνια. Πρέπει λοιπόν να αναλυφθούν πρωτοβουλίες για τις, ε, τους ευρωπαϊκούς πυρνικούς σταθμούς ε, για να προστατευτούμε. Υπάρχουν πολύ σοβαρά γεγονότα και στη Λιβύη. Και εκεί ε, οφείλουμε να ε, συνδράμουμε τον πληθυσμό, να είμαστε έτοιμοι ε, και θα δώσω το λόγο τώρα εις ε, τον εισηγητή κύριο Γκιόρενς, ο οποίος θα ασχοληθεί με αυτό μετά έχετε να κάνετε ανακοινώσεις ε, από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ναι, ε, θα ήθελα να σας ε, αναφέρω πώς προβλέπουμε να αναδιοργανώσουμε την ΕΦΚΟ. Ελπίζω ότι είμαστε στην τελική ευθεία και ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ψηφίσει το οργανόγραμμα στο τέλος του μηνός και μετά θα μπορέσει να σας το ανακοινώσει. Όσον αφορά πολιτικές πρωτοβουλίες. Η επόμενη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα είναι η έκθεση σχετικά με την αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Accountability and Monitoring. Είναι η συνήθις έκθεση την οποία εκδίδουμε κάθε Απρίλιο σχετικά με το επίπεδο βοηθείας που καταβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη και σήμερα είναι σημαντικό ε, να εξετάσουμε την έκθεση αυτή διότι θα αποτελέσει την ε, βάση για τις ε, σκέψεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Ιούνιο όπως είχε αποφασιστεί πέρυσι. Ευχαριστώ. Λοιπόν, το σημείο 7 τώρα θα συζητήσουμε για το σχέδιο εκθέσεως για το μέλλον της δημοσιονομικής στηρίξεως της υποανάπτυξης χώρες από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι το μέλλον του προϋπολογισμού το οποίο θα επακολουθήσει μετά το καλοκαίρι <clears throat> μία ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί του ιδίου θέματος. Ε, πρέπει να καθοριστεί λοιπόν η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του θέματο αυτού και ο κύριος Γκέρενς είναι ο εισηγητής για την κατά έκθεση και δίνω το λόγο στον κύριο Γκέρενς για να παρουσιάσει την έκθεσή του. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν είναι πρώτη φορά που έχουμε την ευκαιρία να προσεγγίσουμε το θέμα αυτό της δημοσιονομικής στήριξης. Σήμερα σας παρουσιάζω ταυτόχρονα με την ε, προφορική μου έκθεση και μια προσωρινή γραπτή εκδοχή διατύπωση που νομίζω ότι έχει μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες εργασίες. Υπάρχει λοιπόν αυτό το έγγραφο το οποίο τίθεται στη διάθεσή σας. Εγώ προσωπικά είμαι πάντοτε αντίθετο σε ψηφίσματα ή προτάσεις ψηφισμάτων που είναι ιδιαίτερος ε, μακροσκελή. Ε, αλλά είναι τμήμα της ε, κοινοβουλευτικής εργασίας να μπορεί κανείς ε, να ελέγξει ακριβώς το μήκος, την έκταση ενός εγγράφου. Αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο προφορικά θα σας παρουσιάσω πιο ξεκάθαρα το θέμα. Ας ξεκινήσουμε καταρχήν από τα αρνητικά σημεία και θα θυμάστε ότι στην πρώτη μου παρουσίαση είχα δώσω την έμφαση στις ανησυχίες σε σχέση με τη δημοσιονομική στήριξη. Και νομίζω θα πρέπει να κινηθούμε έτσι, γιατί η δημοσιονομική στήριξη δεν την χάνει ομόφωνης αποδοχής στις χώρες μέλη. Και μπορούσα να δώσω την έμφαση σε ορισμένα προβλήματα ε, ε, εκ μέρους των χωρών μελών, ε, μια στάση η οποία από τη μία ε, στηρίζει την ε, παροχή δημοσιονομικής ε, στήριξης από τα Ταμεία Ανάπτυξης και αποδέχονται η Επιτροπή να εκτελέσει, να παράσει αυτή τη δημοσιονομική στήριξη και από την άλλη οι ίδιες αυτές χώρες δεν χορηγούν δημοσιονομική στήριξη στο εσωτερικό τους. Δεν το εφαρμόζουν στο εσωτερικό τους. Νομίζω ότι θα πρέπει να μπορούμε να δείξουμε σε εκείνους που έχουν το δικαίωμα ελέγχου ότι, ότι είμαστε ειλικρινείς και ότι θα πρέπει να φέρουμε, ότι ε, αφήστε φέρουμε την ευθύνη, είμαστε και πάρα πολύ αυστηροί. Νομίζω ότι έτσι μπορούμε να παράσχουμε επαρκή προστασία στο επίπεδο των χωρών μελών και να απομακρύνουμε αυτέ τι αμφισημίε. Δεύτερον, όσον αφορά τη δημοσιονομική στήριξη, όλοι γνωρίζουμε τι σημαίνει κάτι τέτοιο πρόκειται για τα κονδύλια τα οποία δεν περιλαμβάνουν τις εκταμιεύσεις στο πλαίσιο συγκεκριμένων προχρωμάτων, αλλά πρόκειται για κονδύλια τα οποία ε, δίδονται προς τις ε, χώρες ε, αποδέκτες και συνδέονται με την επιβολή αυστηρών όρων. Και πρόκειται για την ε, βοήθεια μέσω της δημοσιονομικής στήριξης, η οποία ε, τίθεται αφιβόλω αυτή τη στιγμή δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις. Και βεβαίως αυτό έχει ένα, έχει ένα κίνδυνο μακροοικονομικής ε, αστάθειας που ισοδυναμεί με ένα κίνδυνο μη συνέχισης επενδύσεων σε βασικούς κοινωνικούς τομείς. Ιδού λοιπόν οι δύο βασικές ανησυχίες οι οποίε οποίες εκφράζουν, ε, συνδέονται ακριβώς με αυτή την προβληματική. Ενώ βεβαίως υπάρχουν και θετικά σημεία. Η δημοσιονομική στήριξη είναι ένα ισχυρό μέσο προώθησης ε, της ε, ανάπτυξης και του δυναμισμού ενδογενούς ανάπτυξης των χωρών αποδεκτριών αυτής της βοήθειας σε σχέση με την εξάλληψη, εξάλληψη της φτώχειας και το κείμενο προβλέπει οι χώρες εταίροι του Νότου να τεθούν σε θέση ακριβώς να ε, εξελιχθούν ήδη ε, σε ε, φορείς που καθορίζουν την εξέλιξή τους, πρωταγωνιστές της εξέλιξή τους. Και αυτός είναι ο ρόλος που θα πρέπει να αναλάβουν οι χώρες εταίροι Τώρα, όσον αφορά τις ανησυχίε και πρέπει να τι αμβλύνουμε σε κάποιο βαθμό, ε, θεωρώ ότι θα πρέπει να προσέξουμε σε μια δυναμική προσέγγιση, η οποία κατά την άποψή μου ε, ε, σε σχέση με τις δωρήθριες χώρες ισοδυναμεί με ένα στίχημα για το μέλλον, για τις αποδέκτριες χώρες είναι ισοδυναμεί με την ευκαιρία να αναλάβουν κάποιες δεσμεύσεις όσον αφορά τη δυνατότητα ελέγχου των δημόσιων οικονομικών και τη δυνατότητα διαχείριση των δημόσιων οικονομικών και πρόκειται επίση για μια δέσμευση εκ μέρου των αποδεκτριών χωρών να χαράξουν ένα μέλο ε, μαζί με την συμμετοχή τη ομάδα των ε, κοινωνία των πολιτών. Ε, και θεωρώ ότι αυτό έχει μια διπλή συνέπεια. Εκείνοι οι οποίοι επομίζονται με την εκτέλεση της ε, δημοσιονομικής, την εφαρμογή της δημοσιονομικής στήριξης, θα πρέπει να προσπαθήσουν ώστε να υπάρξουν ε, εταιρικέ σχέσεις με τις ε, χώρες του Βορρά και την Επιτροπή. Δηλαδή, οι συμφωνίες οι οποίες συνάπτονται μεταξύ Επιτροπής Κομισιών και, αποδεκτριών, και χωρών θα πρέπει να είναι προσιτές από όλους τους βουλευτές αυτές τις συμφωνίες. Δηλαδή εμείς ως ε, Ευρωπαίοι βουλευτές, Ευρωβουλευτές θα πρέπει να είμαστε σε θέση να έχουμε προσέγγιση σε αυτά τα κείμενα ε, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να σκηθεί αποτελεσματικό έλεγχος. Και αυτό είναι σε όφελος της Κομισιόν και σε δικό μας όφελος. Ε, προωθώντας λοιπόν τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και μέσω μιας μεγαλύτερης ε, ε, συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών και του Κοινοβουλίου πιστεύω ότι τα βασικά συστατικά εξασφαλίζουν ώστε να κρατήσουμε αυτό το στίχημα για το μέλλον. Αυτό το στίχημα για το μέλλον το οποίο εκφράζει από ακριβώ αυτή τη δυναμική προσέγγιση να έχει ένα σημαντικό πλεονέκτημα. Εάν ε, μέσα του πακέτου αυτού μπορούμε να επικεντρωθούμε σε μια βελτίωση της δυνατότητας απορρόφησης και της καλύτερης διαχείρισης εκ μέρους των χωρών του Νότου. Και αυτό το λέω γιατί πρόκειται για ένα μοντέλο το οποίο θα μπορούσε ενδεχομένω να αποτύχει ή να επιτύχει και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δυναμική προσέγγιση δεν είναι τίποτα άλλο από το στίχημα για το μέλλον στο πλαίσιο της ε, Ευρωπαϊκής Ευρωπαϊκή Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Κάτι το οποίο βεβαίω ορισμένε χώρε επιτυχάνει και σε άλλε αποτυχάνει. Και αν αποτυχάνει, αυτό θα μπορούσε, η αποτυχία αυτή θα μπορούσε να είναι το αποτέλεσμα σφαλμάτων που διαπράττουν οι χώρε αποδέκτε, αλλά θα μπορούσε επίση να είναι σε συνάρτηση με, ατυχή, με την ατυχή συγκυρία της χρηματοπιστωτικής κρίσης την οποία διανύουμε την εποχή αυτή. Ε, συνεπώς δεν μπορούμε να δώσουμε διδάγματα γιατί κανείς δεν είναι αλάνθαστος. Αλλά μπορούμε από την άλλη πλευρά να μεταφέρουμε τη δική μας εμπειρία και να διαπιστώσουμε ότι θα πρέπει να είμαστε κάπως προσεκτικοί με την, όσον αφορά την εφαρμογή αυτού του εργαλείου. Αυτό προϋποθέτει ότι θα πρέπει επίσης να πράξουμε το ώστε τα μέσα του εσωτερικού ελέγχου να βελτιωθούν στο επίπεδο των δύο εταίρων. Όσον αφορά την δυναμική ε, προσέγγιση, μας επιτρέπει να συμφιλειώσουμε τρόπο την τις ε, λαμφάνωσες αδυναμίες της χώρας αποδέκτριες της ε, ε, στήριξης και από την άλλη να τις οδηγήσουμε στο να οικειοποιηθούν βαθμιαία τα ουσιώδη στοιχεία της ιδέας τους της ανάπτυξης. Και υπό την έννοια αυτή θεωρώ ότι όλοι έχουμε κάθε ενδιαφέρον να ενθαρρύνουμε την Επιτροπή να δώσει προτεραιότητα σε αυτό το δρόμο. Βεβαίως, ορισμένες χώρες αποκλείονται ε, από τη δημοσιονομική στήριξη για λόγω συγκεκριμένων αδυναμίων που εφόσον είναι ιδιαίτερα έντονες δεν είναι δυνατόν να δοθεί αυτή η στήριξη. Και αυτό συνδέεται με δύο προβλήματα. Από τη μία θα πρέπει να γίνει μια κριτική αυστηρή αξιολόγηση όσον αφορά τις αποδέκτηρες χώρες και από την άλλη πλευρά ε, εφόσον πρόκειται για χώρες που ε, έχουν μια δύναμη κυβέρνηση και οι χώρες αυτές πολύ συχνά είναι λιγότερο εξελιγμένες και βεβαίως ο πληθυσμός στην περίπτωση αυτή ποινικοποιείται ε, διπλά ακριβώς λόγω αυτής της δυσμενούς κατάστασης και λόγω ακριβώς των περιορισμένων προοπτικών ε, της δημοσιονομικής στήριξης. Και είναι οι ίδιοι πληθυσμοί των χωρών αυτών που αποκλείονται τελικά. Άρα οι πληθυσμοί αυτοί εχμαλωτίζονται λαμβάνοντας όμοιροι σε συγκεκριμένα με αυτά τα κριτήρια διαφάνειας. Ε, εν πάση περιπτώσει, η δημοσιονομική στήριξη δεν συνεπάγεται μια αλλαγή του ε, κυρίαρχου μοντέλου. Ε, δεν τίθεται να τα βασικά και εκτιμένα. Θα πρέπει να συντρέχουν όλες οι προηγούμενες προϋποθέσεις σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Συνένωση όσον αφορά την ανάπτυξη ε, δεν θα πρέπει να, υπάρξουν, να προσέξουμε σε νέες ε, φόρμουλες όσον αφορά τα ουσιώδη κομμάτια της πολιτικής μας. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ακριβώς ε, τόνισα, ε, έθεσα μάλλον αυτά τα κριτικά σημεία τα οποία βεβαίως είναι πιο περιορισμένα σε σχέση με τα μεγάλα πλεονεκτήματα της δημοσιονομικής ε, στήριξης. Εδώ λοιπόν σε ευχαριστώ και περιμένω τις αντιδράσεις σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ε, ευχαριστούμε πολύ κύριε Γκέρνς για την ε, έκθεση αυτή την οποία κατακτήσετε σχέση με τη δημοσιονομική στήριξη. Ε, είναι αλήθεια ότι τελευταία το ζήτημα της δημοσιονομικής ε, στήριξης ε, καταλαμβάνει ένα κεντρικό χώρο στο πλαίσιο της συζήτηση για τις πολιτικές συνεργασίες και στο πλαίσιο της εργασίας μεταξύ των διαφορών θεσμικών οργάνων. Εμείς σήμερα συζητούμε την έκθεση του κυρίου Γκέρενς και στην προσεχή κοινοβουλευτική συνέλευση ΑΚΕ και Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο στην ε, Βουδαπέστη. Θα συζητήσουμε επίσης μια έκθεση για την ε, δημοσιονομική στήριξη, όπου εγώ είμαι εισηγητής εδώ, και η Κομισιόν ε, προτίθεται να αυξήσει τη διάσταση και, του, και το χώρο της δημοσιονομικής στήριξης στο πλαίσιο της γενικής της, της πολιτικής για τη συνεργασία και συνήθως πρόκειται ένα θέμα το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο της ε, συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών οργάνων και στο επίκεντρο της ε, ε, πολιτικής των αποδεκτριών χωρών. Ο κύριος Γκέρνς είπε ότι πραγματικά υπάρχει μια, γίνεται μια πλατιά συζήτηση και εδώ στο Κοινοβούλιο έχουν παρουσιαστεί και κάποιες ε, εκθέσεις σε σχέση με τις αδυναμίες και τα πλεονεκτήματα της δημοσιονομικής στήριξης ως μορφή συνεργασίας. Είναι σίγουρο ότι η γενική θέση την οποία συμμεριζόμαστε εδώ είναι ότι τα πλεονεκτήματα υπερέχουν των αδυναμιών και ότι οι αδυναμίες στην πραγματικότητα είναι κάποιοι κίνδυνοι που θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε, που είναι λοιπόν αποφεύξιμοι και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να τις αποφύγουμε. Ε, Συμμερίζομαι κατά βάση της, ε, την έκθεση του κ. Γκέρενς και νομίζω ότι κατανοώ τόσο εγώ όσο και η πλειονότητα αυτή τη Επιτροπή ότι δεν θα πρέπει η δημοσιονομική στήριξη να πρέπει να συνδέεται με ε, συγκεκριμένους πολιτικούς ή οικονομικούς ε, κανόνες. Και αυτό βεβαίως σημαίνει ότι θα πρέπει να βασίστε σε έναν πολιτικό διάλογο, πολιτικό διάλογο μεταξύ δωρητών και αποδεκτών και, και ανάμεσα δωρητές και αποδέκτες και στο πλαίσιο του οποίου διαλόγου θα πρέπει να ορίζονται οι προτεραιότητες σε σχέση με τις αποδέκτριες χώρες ε, Πρόκειται λοιπόν για έναν πολιτικό διάλογο, ο οποίος επίσης οδηγεί στην κοινή διατύπωση κριτηρίων αξιολόγησης και σε ένα θεμελιώδες στοιχείο του ώστε η δημοσιονομική στήριξη να μπορέσει να αποβεί αποτελεσματική. Αυτό το ουσιαστικό στοιχείο είναι η θεσμική ενίσχυση των χωρών και η δημιουργία συστημάτων ε, δημόσιας ε, διαχείρισης και διοίκησης, η συμμετοχή ε, της κοινωνίας των πολιτών σε αυτές τις διαδικασίες και ο διοικητικός έλεγχος καθώς και ο κοινοβουλευτικός έλεγχος, κάτι στο οποίο θα αναφερθώ στη συνέχεια. Άρα όχι επιβολή όρων, ε, πολιτικός διάλογος και κατάρτιση μέσω αυτού του διαλόγου, διατύπωση των προτεραιοτήτων και των κριτηρίων αξιολόγηση, καθώς και ενίσχυση της, ε, ε, των θεσμών. Θα ήθελα τώρα να επισημάνω ορισμένες πτυχές που λαμβάνονται υπόψη στην έκθεση αυτή, αλλά θα μπορούσαν ίσως να εμπλουτιστούν περισσότερο με την εισφορά των υπολείπων συναδέλφων αυτής της Επιτροπής. Και θα αναφέρω σχετικά ορισμένα στοιχεία. Καταρχήν, σταδιακή προσέγγιση. Το επεσήμανε άλλο ο κύριος Γκέρνς λέγοντας ότι ίσως ορισμένες από τις ανησυχίες που προκαλεί η δημοσιονομική στήριξη συνδέεται με το γεγονός ότι ξαφνικά ε, θα αλλάξουμε την πολιτική μας συνεργασία και θα περάσουμε στην, σε μια άλλη κατάσταση που επενδύουμε όλες τις προσπάθειες στην δημοσιονομική στήριξη. Αλλά αυτό δεν ισχύει. Πρόκειται για μια σταδιαία διαδικασία ενίσχυσης και παροχής της δημοσιονομικής στήριξης. Και αυτή η σταδιαία ε, η σταδιακή παροχή στήριξης συνδέεται ακριβώς με τη θεσμική ενίσχυση των χωρών που αποδέχονται τη στήριξη αυτή. Κατά δεύτερο λόγο, θα ήθελα να αναφερθώ συμβατότητα, το οποίο σημαίνει ότι η δημοσιονομική στήριξη δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να αντικαταστήσει άλλους τρόπους στήριξης. Δεν πρόκειται να βάλει στην άκρη άλλες μορφές ε, βοήθειας, αλλά θα πρέπει να καταστεί συμβατή ακριβώς με τις άλλες μορφές βοήθειας και θα πρέπει ακριβώς ε, να υπάρξει προσπάθεια τους να υπάρξει ένας καλύτερος εσωτερικός συντονισμός μεταξύ των διαφόρων μορφών ε, παροχής βοήθειας. Τρίτον, ο κύριος Γκέρενς είπε ότι δεν είναι λογικό στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέσω της Επιτροπής να έχουμε μια πολιτική επέκταση της δημοσιονομικής στήριξης ε, σε σχέση με συγκεκριμένα κριτήρια, ενώ οι χώρες μέλη αγνούν αυτές τις αρχές. Κάτι τέτοιο δεν είναι σωστό. Τέταρτον, και εδώ θα κλείσω, διατύπωση προτεραιοτήτων. Αυτό σημαίνει ότι παρόλο που οι χώρες που αποδέχονται τη στήριξη ε, λειτουργούν σύμφωνα με τη βασική αρχή ε, οικειοποίηση τη δυνατότητα να ορίζουν μόνε του οι χώρε αυτέ τι δικέ του προτεραιότητε, θα πρέπει να υπάρξει ένα διάλογο ώστε να καταλήξουμε ε, στο συμπέρασμα η εκπαίδευση και η εξάλληψη της ε, φτώχειας να ε, γίνουν οι βασικές ε, προτεραιότητες και προϋποθέσεις της δημοσιονομικής στήριξης. Τέλος, θα ήθελα να πω ότι με τον ίδιο τρόπο προσπαθούμε εδώ να παίξουμε ένα πιο αποφασιστικό ρόλο σε Ευρωβουλή στα πλαίσια της πολιτικής συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε τα εθνικά κοινοβούλια των χωρών που είναι αποδέκτες της στήριξης αυτής να μπορέσουν να ορίσουν μόνες τους τις δικές τους προτεραιότητες ορίζοντας ακριβώς ε, τα κριτήρια και ασκώντας ε, κοινοβουλευτικό έλεγχο. Στο βαθμό αυτό θα ήθελα να πω ότι στηρίζω την έκθεση του κυρίου Γκέρενς. Ευχαριστώ πολύ. Merci beaucoup. Ευχαριστώ. Νόησα. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος. Η έκθεση του συναδέλφου Γκιόρενς είναι καλή, είναι καλή και από πλευράς περιεχομένου και επίσης παρουσιάζεται πολύ έξυπνα διότι λαμβάνει υπόψη τις ανησυχίες των κρατών μελών και πολλών ευρωβουλευτών. Νομίζω ότι στον τομέα της δημοσιονομικής βοηθείας πρέπει ε, να διευκρινίσουμε πολλά θέματα προς τους συναδέλφους, ιδίως όταν μιλάμε με συναδέλφους της Επιτροπής Προπολογισμού διαπιστώνουμε ότι εκεί υπάρχουν πολλές επιφυλάξεις για την δημοσιονομική βοήθεια. Εγώ θέλω να αναφερθώ ουσιαστικά σε δύο θέματα, διότι στο σημείο 5 ο κύριος Γκέρενς μιλά για την κοινωνία των πολιτών και για τα εθνικά κοινοβούλια που θα πρέπει να συμμετέχουν στις διαβουλεύσεις και αυτή τη στιγμή ε, προσπαθούμε να ολοκληρώσουμε τον ε, σωστά οργανωμένο διάλογο όπου συμμετέχουν και οργανώσεις που πρέπει να συμμετάσχουν πέραν των, της κοινωνίας των πολιτών και των εθνικών κοινοβουλίων. Στο σημείο 14 επίσης ο κύριος Γκιόρενς γράφει ότι πρέπει να πιέσουμε για τον συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να υπάρξει μια βελτίωση διότι διαπιστώνουμε ε, στην εξωτερική πολιτική ότι δεν υπάρχει κοινή αντιμετώπιση τουλάχιστον στο θέμα της Λιβύης παραδείγματος χάρη. Θα πρέπει να υπάρξει ένας καλύτερος συντονισμός μεταξύ κρατών μελών και Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και ε, μεταξύ μας. Τέλος, ο συνάδελφος Ενρίγε Γκερέρο είπε ότι όλα αυτά μπορεί να γίνουν μόνο σε ένα πλαίσιο διαλόγου. Αλλά μπορούμε να απαιτήσουμε και κάτι παραπάνω. Μπορούμε να το συνδυάσουμε με προϋποθέσεις για την δημοσιονομική βοήθεια και ε, για να μπορέσουμε ε, να καταρτήσουμε δομές όπου θα πούμε ότι η δημοσιονομική στήριξη θα προωθήσει τα ανθρώπινα δικαιώματα, θα πρέπει να διαπιστώνουμε ότι υπάρχει εκδημοκρατισμός. Θα πρέπει να πούμε ότι έχουμε ένα ελεγκτικό συμβούλιο το οποίο ελέγχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ολοκληρώνοντας όμως ευχαριστώ τον κύριο Γκέρενς για την ε, έκθεσή του και για την παράθεση των ανησυχιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην αρχή και την πρόθεσή του να συμμετάσχει και η κοινωνία των πολιτών. Θα ήθελα να καλωσορίσω και την ομάδα επισκεπτών του κυρίου Γκέρενς από το Λουξεμβούργο. Μπέρμαν. Να καλωσορίσω και εγώ τους Λουξεμβούργιους επισκέπτες. Ήρθατε να μας δείτε στο φυσικό μας περιβάλλον κάποιες παρατηρήσεις για τη δημοσιονομική στήριξη. Είμαι εισηγητή στην Επιτροπή Προϋπολογισμού για το συγκεκριμένο θέμα και καταλήγουμε στην έκθεσή μας σήμερα επί τη βάση της εκθέσεως ε, του ελεγκτικού συνεδρίου. Η έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου ασκεί οξία κριτική στην πολιτική που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη Δημοσιονομική Στήριξη. Τα ευρήματα του συνεδρίου δείχνουν ότι οι κίνδυνοι δεν αντιμετωπίζονται σωστά στα πλαίσια των διαδικασιών τις οποίες χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δύο είναι οι κίνδυνοι. Πρώτον, ότι τα χρήματα καταλήγουν στις λάθος τσέπες Υπάρχει εδώ θέμα κατάχρησης. Και το δεύτερο είναι να χρησιμοποιηθούν για τα προγράμματα αυτά τα χρήματα, αλλά να μην παράγουν τα αποτελέσματα τα αναμενόμενα. Και αυτά είναι πράγματα που πρέπει να αλλάξουν. Οι διαδικασίες θα πρέπει να συμπεριλάβουν μετρήσιμους δείκτες, οι οποίοι θα πρέπει να είναι ποσοτικοποιήσιμοι και τότε μόνο θα μπορούμε να μπούμε ότι η δημοσιονομική στήριξη έχει πραγματικά ε, ουσιαστικά αποτελέσματα. Ταυτόχρονα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιμετωπίζει το θέμα με δυναμικό τρόπο. Για να είναι επιλέξιμο ε, ένα κράτος για δημοσιονομική στήριξη πρέπει να επιδεικνύει ένα κάποιο επίπεδο καλής διακυβέρνησης, υγιούς δημοσιονομικής πολιτικής και διαχειριστικής πολιτικής κτλ. Αυτά έχουν σημασία βέβαια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί επίσης ότι ορισμένες χώρες ε, οδεύουν προς χρηστή διακυβέρνηση και καλύτερη οικονομική διαχείριση των ε, δημοσιονομικών τους. Και αυτές οι χώρες οι οποίες είναι ε, προς τον στόχο αυτό θα πρέπει να είναι και αυτές επιλέξιμες. Τίθεται λοιπόν το θέμα εδώ ότι από τις 30 χώρες που παίρνουν δημοσιονομική στήριξη σήμερα, 12 δείχνουν εξαιρετικά άσχημα αποτελέσματα στον δίκτυο διαφθοράς. Κάτω από το 3 με ανώτερο το 10. Εφόσον ισχύει κάτι τέτοιο και εφόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι ο γενικός προϋπολογισμός είναι το σωστό μέτρο, τότε θα πρέπει να υπάρξουν μέθοδοι παρακολούθησης ιδιαίτερα διαφανείς και αποτελεσματική, και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει αρκετό προσωπικό στις αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν ξεκινήσουν οι διαδικασίες αυτές που μπορεί να οδηγήσουν σε πραγματικούς κινδύνους σε επίπεδο εμπιστοσύνης. Υπάρχουν και άλλα θέματα εδώ. Προφανώς και απαιτείται ένας σωστός πολιτικός διάλογος με την χώρα αποδέκτη. Ε, δεν στηρίζουμε ένα συγκεκριμένο προϊόν, δεν συγκρίνουμε μια πολύ απλή μορφή αναπτυξιακής βοήθειας. Η γενική ε, δημοσιονομική στήριξη δίνει τη δυνατότητα να ενταχθεί κανείς σε ένα στενό πολιτικό διάλογο με τις χώρες αποδέκτες και τις κυβερνήσεις τους. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρξει ισχυρή πολιτική βούληση και αποφασιστικότητα ο τρόπο αντιμετώπισης του θέματος από όλα τα κράτη-μέλη και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί τότε μόνο μπορεί να επωφεληθεί κανείς από την προστιθέμενη αξία των 27 συν την Επιτροπή και από το πιθανό πολιτικό βάρος το οποίο ε, συνεπάγεται. Όταν είμαστε ενωμένοι μπορούμε να παίξουμε ένα ισχυρό πολιτικό ρόλο. Βέβαια δεν είναι εύκολο να συμβεί κάτι τέτοιο. Τα κράτη-μέλη κάνουν ό,τι θεωρούν καλύτερο, δυσκολεύονται να συντονίσουν ε, όταν δεν το επιθυμούν αυτό, όταν δεν θεωρούν ότι πρέπει να λειτουργήσουν συντονισμένα. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αλλάξει εφόσον η δημοσιονομική στήριξη θα πρέπει να καταστεί το αποτελεσματικό μέσο που θα θέλαμε. Συμφωνώ με αυτά που είπε ο Γκέρενς ότι είναι πολύτιμο το μέσο αυτό δυνητικά ε, γιατί βοηθά θα έλεγα την ευαισθητοποίηση των κυβερνήσεων αποδεκτών και ενισχύει γενικότερα και τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών. Είναι σημαντικά όλα αυτά, αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες οι οποίοι παίζουν εδώ ένα συγκεκριμένο ρόλο πριν γίνει η βοήθεια αυτή μέσω της δημοσιονομικής στήριξης πραγματικά πολύτιμη. Ευχαριστώ Λεβίν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον κύριο Γκέρενς για την έκθεσή του. Δεν είμαι εμπειρογνώμων στα θέματα δημοσιονομικής στήριξης, άκουσα όμως τη συζήτηση η οποία παρουσιάζει πολύ ενδιαφέρον. Συμφωνώ με τις ανησυχίες τις οποίες εξέφρασε ο Μπέρμαν. και νομίζω ότι ανάμεσα σε αυτά τα οποία είπε ο κύριος Γκέρενς ε, υπάρχουν πολλά τα οποία προκαλούν ερωτηματικά. Καταρχάς, οι συνθήκες που επιβάλλονται στις χώρες οι οποίες είναι επιλέξιμες για δημοσιονομική στήριξη. Πρέπει να υπάρξουν όροι και προϋποθέσεις για τη βοήθεια αυτή. Οι προϋποθέσεις αυτές όμως θα πρέπει να είναι συμβατή με τις αρχές και τους κανόνες που έχει θέσει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Παγκόσμια Τράπεζα για την απελευθέρωση των αγορών, τη διαχείριση των εθνικών πόρων κτλ. Εφόσον είναι ένα από τα κριτήρια, αυτό είναι κάτι λοιπόν το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει. Τώρα το θέμα της διαφάνειας αν τα χρήματα πηγαίνουν απευθείας στον γενικό προϋπολογισμό των χωρών αποδεκτών, έχουμε ένα θέμα διαφάνειας, από ό,τι γνωρίζω, στα πλαίσια της συζήτησης αυτής και ανάμεσα ε, στις κριτικές που ακούονται ε, προς την ε, δημοσιονομική στήριξη, υπάρχει το λεγόμενο παρασιτικό φαινόμενο, δηλαδή όταν πηγαίνουν κάποια χρήματα σε γενικούς τομείς όπως η παιδεία, όπως η υγεία κτλ. Δημιουργείται ένας οικονομικός χώρος για την κυβέρνηση να χρησιμοποιήσει τα χρήματα αυτά και για στρατιωτικούς σαν παράδειγμα λόγους. Δεν θα θέλαμε να συμβεί κάτι τέτοιο. Αυτό λοιπόν το φαινόμενο του παρασιτισμού είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί όταν μεταφέρονται οι δημοσιονομικά μέσα προς τις χώρες αυτές και το θέμα της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών, της συμμετοχής των κοινοβουλίων στις συζητήσεις με τις χώρες αποδέκτριες είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα εφόσον θέλουμε οι χώρες να αποφύγουν αυτήν την τεράστια δυνατότητα διαφθοράς και πολλές θυμίζω από τις χώρες όπως είπε ο κύριος Μπέρμαν που παίρνουν τέτοια χρήματα στα πλαίσια της δημοσιονομικής στήριξης είναι πολύ χαμηλά τον δείκτη διαφθοράς ή πολύ ψηλά όπως θέλετε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ο Τσάρλς Γκάρενς ως συνήθως έχει κάνει εξαιρετική εργασία ε, επί ενός πολύ περιορισμένου θέματος ιδίως από ό,τι εμείς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουμε κάνει σχετικά με τη δημοσιονομική στήριξη. Σαν Επιτροπή όμως κυρία Πρόεδρε, η οποία εποπτεύει τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, πρέπει να επιμείνουμε τώρα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να έρχεται και να μας λέει τι έχει δαπανίσει, αλλά τι έχει δαπανίσει και ε, τι απέδωσε η δαπάνη αυτή. Ξέρω ότι στην προηγούμενη συνεδρίαση είχαμε πει πόσο δύσκολο είναι ε, να αλλάξει κανείς τις δομές του και για να μετρήσει το αποτέλεσμα και να δεσμευτεί για αποτέλεσμα, αλλά όταν μιλάμε για 29 εκατομμύρια δαπάνες παραδείγματος χάρη σε προγράμματα χωρών, ε, όταν τους ρωτήσετε πόσα νοσοκομεία χτίστηκαν, πόσα παιδιά παιδιά εκπαιδεύτηκαν, πόσοι ασθενείς θεραπεύτηκαν, δεν ξέρουν. Στα πλαίσια λοιπόν της ε, δημοσιονομικής στήριξης αυτό είναι μια πολύ νοχέλικη ε, εξέλιξη. Δίνετε τα χρήματα και γεια σας. Δεν είναι έτσι, δεν είναι ο σωστός τρόπος για να χρησιμοποιούμε τα χρήματα των ε, πολιτών και των φορολογουμένων μέχρι ότου λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορέσει να μετρήσει το αποτέλεσμα θα πρέπει να γίνουμε πολύ ε, επιφυλακτικοί ε, για το τι θα κάνουμε με την δημοσιονομική στήριξη. Μετά υπάρχει και ένα άλλο θέμα Ορισμένες χώρες είναι φτωχές, όχι γιατί δεν έχουν χρήματα, όπως η Νιγηρία παραδείγματος χάρη, αλλά διότι δεν έχουν τις τεχνικές ικανότητες, το κατάλληλο, τους κατάλληλους δημοσίους υπαλλήλους, τα στελέχη, τις συμφωνίες και ούτω καθεξής. Άρα το να δώσει κανείς χρήματα στις υποανάπτυξη χώρες προϋποθέτει ότι ο λόγος για τον οποίο είναι φτωχές είναι διότι δεν έχουν χρήματα λάθος. Δεν ξέρουν πώς να διαχειριστούν τα προβλήματα της οικονομίας τους και γι' αυτό είναι φτωχές. Δεν ξέρουν πώς να προκαλέσουν ο πλούτο, πώς ε, θα ε, μπορέσουν να έχουν μια ανταγωνιστική οικονομία. Και ε, βάσει της ε, και έτσι εάν δίνουμε δημοσιονομική στήριξη είμαστε τεμπέληδες και δεν βοηθούμε στο να αναπτύξει κανείς τις ικανότητες αυτές. Επιπλέον μπορεί να υπάρξει τεράστια ε, διαφθορά διότι η τεχνολογία και η μεθοδολογία δεν υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ελέγξουν την ύπαρξη ή όχι διαφθοράς. Υπάρχει και μεταφορά. Αν είμαι μια χώρα η οποία θέλει να δαπανίσει χ στις υγειονομικές υπηρεσίες και Ψή ή ε, τις αμυντικές μου δαπάνες για να αγοράσω τάγκς, ε, όπλα και αεροπλάνα. Δεν έχω χρήματα διότι θα πρέπει να χρηματοδοτήσω τα νοσοκομεία ή την παιδεία. Έρχεται λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση και μας λέει σας δίνουμε 30 εκατομμύρια για σχολίδια ή νοσοκομεία. Οπότε ε, λέω θαυμάσια, αλλά ε, βάζω τα χρήματα αυτά εις ε, τα σχολεία και στα νοσοκομεία, αφαιρώ όμως από τον εθνικό προϋπολογισμό το αντίστοιχο κεφάλαιο και αγοράζω οπλισμούς. Αυτό πώς θα το σταματήσουμε. Ακόμη και αν υπάρχει ένα σωστό ο λογιστικό σύστημα και εποπτικό σύστημα το οποίο παρακολουθεί ε, το, την ε, εφαρμογή του εθνικού προπολογισμού και τις ε, δικές μας προσφορές δεν προχωράμε διότι δεν υπάρχει αρκετή διαφάνεια κατά τρόπον ώστε όπως εμείς θεωρούμε σαν ισότιμου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να γίνει αυτό το οποίο γίνεται ε, σε μια κυβέρνηση να μπορεί δηλαδή ο κάθε βουλευτής να αμφισβητήσει τον ηθικό χαρακτήρα και την τιμιότητα. Τον ε, λόγο έχει ο ο κύριος ε, Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, ε, πιστεύω ότι είναι σωστή η παρουσίαση της ε, εκθεσής αλλά δεν εμφανίζεται σωστά ο, ο αποκεντρωτισμός διότι ε, υπάρχουν συχνά τελευταίως διάφορα θέματα δηλαδή η διαπίστωση ότι οι δαπάνες δεν δεν φτάνουν μέχρι το τοπικό επίπεδο για να μπορέσουν να συνδράμουν την εδαφική εξέλιξη που είναι ανεξάρτητη για μια σωστή ανάπτυξη και από αυτή την σκοπιά οι τοπικές ε, αρχές ε, πρέπει να παίξουν το ρόλο τους, είναι επιτόπου, γνωρίζουν τις ανάγκες ε, των κοινοτήτων τους, είναι αρμόδιες από πλευράς εκπαιδεύσεως, εξυγιάνσεως, υγιεινής κτλ. Πιστεύω λοιπόν ότι μία τομεακή και τοπική κατανομή πρέπει να υπάρξει στις υποανάπτυξη χώρες και γι' αυτό θα προτείνω μία τροπολογία επ' αυτού του θέματος ή στον εισηγητή, ο κύριος Ματίνες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα πρωτίστως να συγχαρώ τον κύριο Γκέρες γιατί ε, όπως τον συνεχάρει και ο κύριος ε, Ντέβα από τα δεξιά εγώ θα, την, θα τον συγχαρώ από τα αριστερά και ε, βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει ένα ευρύ φάσμα στήριξης από δεξιά και από αριστερά για την έκθεση αυτή. Νομίζω ότι εστιάζει σε ένα θέμα το οποίο τίθεται στη συζήτηση εδώ και πολλές δεκαετίες. Δεν μπορούμε να προσθέσουμε πολλά περισσότερα σε αυτά τα οποία είπαν οι συνάδελφοι. Εγώ απλώς θέλω να πω ότι είμαι υπέρ της δημοσιονομικής στήριξης, παρόλο που καταλαμβάνω τους ε, κινδύνους που εξαγγέλθηκαν εδώ και 40 χρόνια όταν, ε, για παράδειγμα, ένα βρέφος ε, συνηθίζει το μπιμπερό και αρνείται άλλους τρόπους λήψης τροφής, τελικά μπορεί να πεθάνει. Πρόκειται λοιπόν για αυτό το φαινόμενο το οποίο μας απειλεί εδώ. Και εάν ε, ε, και υπάρχουν χώρες οι οποίες τελικά αρνούνται να αναπτύξουν μηχανισμούς αυτοδιάθεσης τελικά και ανάπτυξης του δικού τους δυναμικού και αρκούνται σε αυτή την ε, ε, τροφοδοσία από την δημοσιονομική στήριξη. Λοιπόν, θα πρέπει, δεν θα πρέπει να είναι αυτή η δική μας φιλοδοξία, η φιλοδοξία των αποδεκτρών χωρών, δηλαδή να θυστούν στο να επιβιώνουν στη βάση της δημοσιονομικής στήριξης που δέχονται εκ των έξωθεν. Έξωθεν, συγγνώμη. Ε, όπως είπε και η κυρία Λέβιν, θα ήθελα να πω ότι ενισχώ για το γεγονός ότι ε, μεταξύ των κριτηρίων αναφέρεται η ανάγκη ε, προσαρμογής σε καταστάσεις που έχει επιβάλει, για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Και το τελευταίο σχόλιο το οποίο θα ήθελα να κάνω με οδηγεί στο παράδοξο το οποίο έχουμε ζήσει εμείς εδώ ε, εδώ και κάποια χρόνια προσπαθώντας να πετύχουμε όλα τα προγράμματα συνεργασίες ε, να έχουν σαν αποτέλεσμα τελικά οι αποδέκτερες χώρες να μπορούν να ορίσουν τις δικές τους προτεραιότητες. Και η πραγματικότητα είναι ότι έχουμε αντιμετωπίσει το εξή παράδοξο, ότι όταν ε, οι χώρες προσπαθώντας να ασκήσουν τη δική τους αρχή αυτοδιάθεσης και κυριαρχία, όταν οι δικές τους προτεραιότητες δεν συμπίπτουν με τις δικές μας ή με αυτές που τελικά θεωρούμε ότι είναι οι δικές μας προτεραιότητες, τελικά θέτουμε ένα αμφιβόλο αυτή την βασική αρχή ότι θα πρέπει να είναι οι ίδιες οι χώρες που θα πρέπει να ορίζουν τις προτεραιότητες κλπ. Άρα λοιπόν θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αναζητήσουμε κάποιες λύσεις μέσω του διαλόγου και να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε ποιες είναι οι προτεραιότητες των χωρών αυτών και ε, να δούμε ε, και ποιες είναι οι απαιτήσει των δικών μας ε, πολιτών από την άλλη. Ενρικε, σε σχέση με τρία ή τέσσερα σημεία που αφορούν την εκπαίδευση, την υγεία, την εξάλληψη της φτώχειας, αναφέρθηκε σε αυτές ολοκληρώνες, αλλά νομίζω ότι η τεσσερα σημεια που αφορουν την εκπαιδευση την υγεια την εξαλληψη της φτωχειας αναφερθηκε σε αυτες ολοκληρωνες αλλα νομιζω οτι η να πεις κάτι το οποίο είναι θεμελιώδες και που είναι ακριβώς η βοήθεια σε μια γεωργία, γεωργική οικονομία βιώσιμη, επιβίωσης. Ε, βλέπουμε για παράδειγμα στο πλαίσιο της ΑΚΕ, όταν ε, βλέπουμε τις προτεραιότητες που παρουσιάζουν οι διάφορες ε, χώρες εταίροι μας, καμιά από αυτές τις χώρες στην ουσία δεν εισάγει το στοιχείο ακριβώς της γεωργίας επιβίωσης. Ενώ στην πραγματικότητα όλοι διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μια τρομακτική επιδίνωση του ιδίου ε, του παραγωγικού δυναμικού. Ε, γι' αυτό λοιπόν έχω την εντύπωση ότι και αυτό θα πρέπει να αποτελέσει ένα ε, θέμα προτεραιότητας το οποίο θα πρέπει να συμπεριληφθεί εδώ όταν λέμε στους ανθρώπους ότι η υγεία και η εκπαίδευση είναι σημαντικές κλπ. Θα πρέπει να πούμε ότι και αυτό το στοιχείο είναι ιδιαίτερο σημαντικό, δηλαδή η δυνατότητα να παράγει μια χώρα γεωργικά προϊόντα τα οποία να τους επιτρέπει να επιβιώνουν. Θεωρώ ότι είναι μια σημαντική προτεραιότητα. Αυτό είναι το οποίο ήθελα να πω κυρία Πρόεδρε και σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος ε, Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ξεκινήσω ευχαριστώντας τον συγκητή τον κύριο Γκέρες για την εκθεσία του και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική λόγω ακριβώς της βαρύτητας της δημοσιονομικής στήριξης. Και θα ήθελα να επισημάνω ορισμένα από τα πλεονεκτήματα της δημοσιονομικής στήριξης που ανέφεραν και άλλοι συνάδελφοι άλλωστε σε σχέση ακριβώς με την αποτελεσματικότητα αυτής της ε, στήριξης. Πρωτίστως η αρχή της ε, διατύπωσης των προτεραιτήτων εκ μέρους των χωρών αυτών και της οικειοποίησης, της δυνατότητας εξοποίησης του δικού τους δυναμικού ούτε ώστε οι αναπτυσσόμενε χώρε να μπορέσουν να εκφράσουν τι δικέ του ανάγκε στο πλαίσιο του διαλόγου. Δεύτερον, θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν οι εισφορές των δωρητών με τις προτεραιότητες που διατυπώνουν οι αποδέκτες χώρες. Αλλά ίσως ένα από τα σημαντικά ζητήματα και που συμμερίζονται πολλά μέλη αυτής της Επιτροπής είναι η ανάγκη να ενισχύσουμε τους μηχανισμούς κοινοβουλευτικού ελέγχου και τον εποπτικό έλεγχο ε, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ε, το στοιχείο αυτό στο πλαίσιο της ε, δημοσιονομικής στήριξης. Τώρα το λόγο έχει ο κύριος ε, Χωσέ Κορέρα Μουνές εκ μέρους της Επιτροπής και θα ήθελα παρακαλώ να σας παρακαλέσω να είστε σύντομος ούτως ώστε ο κύριος Κέρνς να μπορέσει και αυτός να απαντήσει. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος γιατί το διάλογο αυτό το κάνουμε εδώ και κάποιους ε, μήνες. Ήδη αυτή τη στιγμή ε, ξεκινήσαμε τις εργασίες μας, ο διάλογος αυτός ε, απεδείχθη ιδιαίτερος καρποφόρος και μας επέτρεψε στο πλαίσιο της Πράσινης Βίβλου να συμπεριλάβουμε κάποιες ιδιαίτερες σημαντικές συστάσεις για ορισμένα θέματα τα οποία τίθενται στο πλαίσιο της Πράσινης Βίβλου και όπως είπατε και εσείς, αυτή τη στιγμή επεξεργαζόμαστε τη σύνταξη μιας ανακοίνωσης για τη δημοσιονομική στήριξη και συνεπώς οι συζητήσεις αυτές θα τροφοδοτήσουν και τους δικούς μας προβληματισμούς δεν θα μακρηγορήσω, έλαβα γνώση των δικών σας συστάσεων στο πλαίσιο της συζήτησης, αλλά θα ήθελα παρόλα αυτά να υπογράψω δύο-τρία σημεία. Το πρώτο σημείο αφορά ε, την ε, διατύπωση κάποιων όρων και το ζήτημα της εθνικής ευθύνης. Ε, είναι κάτι το οποίο ήταν ιδιαίτερα έντονο στι διαβουλεύσει για την Πράσινη Βίβλο. Και θα ήθελα να σα πω ότι αυτό είναι ένα θέμα στο οποίο έχουμε εμβαθύνει στο πλαίσιο των υποεξέλιξη εργασιών και υπάρχουν ενδείξει ότι ο Επίτροπο κ. Πίλμπαξ ε, ε, διατύπωσε απόψει σε σχέση με το θέμα αυτό που δείχνουν ότι η Επιτροπή προσπαθεί πράγματι σοβαρά να συμπεριλάβει αυτά τα στοιχεία. Το ίδιο ισχύει και το ζήτημα τη διαφθορά. Είδα ότι συζήτηση, ότι συζήτηση εδώ υπήρξαν κάποιες ε, τοποθετήσεις που εντάσσονται στο πλαίσιο των εργασιών που εξελίσσουμε στο πλαίσιο ακριβώ τη ανακοίνωσή μας. Υπήρξαν κάποιες άλλες ε, παρεμβάσεις που σχετίζονται με τη διαπίστωση που κάναμε και εμεί οι ίδιοι για την αδυναμία του συστήματο και τη διαπίστωση που έκανε και το Ελεγκτικό Συνέδριο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αλλά όταν συζητούμε ζητήματα διαφθορά και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θέτει η πράσινη βίβλο και στο οποίο θα εμβαθύνει και η δική μα ανακοίνωση, θα πρέπει να πούμε ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερο σύνθετο θέμα. Όταν μιλούμε για κάποιου δείκτε, για παράδειγμα, αυτή στιγμή εργαζόμαστε με κάποιου τέτοιου δείκτε. Θα πρέπει να δούμε ποια είναι η συστοιχία, η συνάφεια των διαφόρων όρων δικτών με τη διακυβέρνηση. Και εδώ βλέπουμε ότι δεν υπάρχει μια, ένας ιδιαίτερος έντονο συσχετισμό συνάφεια. Για παράδειγμα στην Κένια, που είναι μια χώρα όπου, επίπεδο, όπου το επίπεδο της ε, είναι ε, ιδιαίτερος υψηλό. Αλλά εάν δούμε τους δείκτες δημοσιονομικής διαφάνειας, βλέπουμε ότι η Κένια βρίσκεται σε μια λογική θέση, δηλαδή κάτω από το μεσό όρο. Ε, πάνω από το μεσό όρο, συγγνώμη. Αυτά είναι στοιχεία λοιπόν τα οποία θα πρέπει να λάβουμε υπόψη, αλλά μπορώ να σα πω ότι εδώ πρόκειται για ένα τομέα που, που εργαζόμαστε ήδη και κοιτάμε τα πράγματα εκ του σύνεγγυ. Τώρα, όσον αφορά τα αποτελέσματα, εάν υπάρχει μια οργάνωση η οποία ε, ασχολείται με την προσέγγιση αυτή, είναι η ίδια η Επιτροπή. Μια προσέγγιση που βασίζεται ακριβώ στα αποτελέσματα. Αυτή είναι η προσέγγιση τη Επιτροπή. Αλλά βεβαίω εδώ υπάρχουν ορισμένε δυσκολίε στο να δούμε ποια είναι αυτά τα αποτελέσματα. Ε, οι άλλοι οργανισμοί, η Αφρικανική Τράπεζα Επενδύσεων, η Κεντρική Τράπεζα κλπ. προσπαθούν να βελτιώσουν τι δικέ του ε, προσεγγίσει. Η, η Κεντρική Τράπεζα ζήτησε να μα δει γιατί ξέρει ότι δουλεύουμε ε, πάνω στα θέματα αυτά. Και ε, γίνεται μια προσπάθεια να βελτιωθεί μια προσέγγιση η οποία να βασίζεται ακριβώ στην επίτευξη αποτελεσμάτων. Αλλά και ίδια η προσέγγιση βασίζεται σε αποτελέσματα που εισήχθησαν το 2000 στην ανακοίνωση, μέσω της ανακοίνωσης της Επιτροπής. Τώρα, το τελευταίο σημείο το οποίο θα ήθελα παρόλο θα υπογραμμίσω είναι η σχέση της Επιτροπής με τις χώρες μέλη. Θα πρέπει εδώ να ξεχνάμε ότι εγκαιτέρως μετά την ανακοίνωση του 2000, ο συντονισμός επιτόπου με τις χώρες ε, μέλη έχει ενισχυθεί. Η δημοσιονομική στήριξη στις περισσότερες χώρες, ιδιαίτερως εκεί όπου υπάρχουν άλλα εμπόδια, γίνεται μέσω ε, έντονων ε, ισχυρών μηχανισμών συντονισμού. Και η Επιτροπή καθώς και χώρες μέλη ήδη από τον περασμένο χρόνο σύστησαν μια ομάδα εργασίες μια ομάδα εργασίες για να ενισχυθεί ακριβώς ο συντονισμός όσον αφορά τη δημοσιονομική στήριξη. Και μπορώ να σας βεβαιώσω ότι έστω και αν στην αρχή οι συζητήσεις ήταν πολύ έντονες και υπήρχαν πολλές αποκλήξεις απόψεων, βαθμιαία εγκαθιδρύθηκε ένα κλίμα εμπιστοσύνης και βλέπουμε ενδιαφέρονται κάποια αποτελέσματα. Άρα λοιπόν ο συντονισμός έχει βελτιωθεί αισθητά και ελπίζουμε ότι μετά την ανακοίνωση αυτή θα μπορέσουμε να υποβάλουμε συγκεκριμένε ε, προτάσεις οι οποίες θα εγκριθούν από το Συμβούλιο ήδη αυτό το χρόνο ή στις αρχές του επόμενου έτους. Τώρα το λόγο έχει ο κύριος Γκέρενς. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Γκερέρο, ο οποίος είναι υπεύθυνο για την Επιτροπή ΑΚΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα πρέπει να παρουσιάσουμε μια ιδέα στην οποία συμμερίζονται συνάδελφοι και ε, δεν πρέπει κανείς να ε, υποτιμήσει τις κριτικές που απευθύνουμε διότι ε, νομίζω ότι η γνώμη πρέπει να καθησυχαστεί όσον αφορά την δημοσιονομική στήριξη. Συμφωνείτε, βλέπω ότι πρέπει να υπάρξουν έξυπνες ε, λύσεις. Ε, ε, νομίζω ότι δεν είναι αξιολόγηση λανθασμένη όταν λέμε ότι εδώ και 30 χρόνια παράγουμε ακριβώς ε, την ίδια ποσότητα των ο, τροφίμων ανακεφαλήν ε, εκτός από ε, το, ότι στο Σαχέλ τριπλασιάστηκε ο πληθυσμός τα τελευταία 30 χρόνια, άρα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι θα πρέπει να υπάρξουν τριπλασιασμοί επίσης παραγωγής. Η κυρία Λαβίν έχει ε, δίκιο όταν ε, ε, κάνει τα σχολιά της, διότι εγώ πιστεύω ότι δεν μπορούμε να βασιστούμε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και στην Παγκόσμια Τράπεζα, γιατί και αυτοί μπορούν να κάνουν λάθος. Και νομίζω ότι εάν οι υποανάπτυκτες χώρες, όλες οι αναπτυγμένες χώρες είχαν όλες καλύψει το 0,7% η κατάσταση στις υποανάπτυξη χώρες θα ήταν τελείως διαφορετική. Μπορεί να κάνει όπως είπα λάθος και η Παγκόσμια Τράπεζα διότι βλέπουμε ότι όσες ε, χώρες προχώρησαν ε, σε αλλαγές χωρίς να λάβουν υπόψη τις αποφάσεις της ε, και τις αξιολογήσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας πήγαν καλύτερα από ό,τι άλλες. Ε, είμαστε όμως οι πρώτοι δανειοδότες. Γιατί να είμαστε ε, τόσο μετριόφρονες. Δεν πρέπει εμείς ε, να ευθυγραμμιστούμε στις αποφάσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ή της Παγκοσμίου Τραπέζης. Εμείς σαν πρώτοι δανειοδότες πρέπει να χαράξουμε τη γραμμή. Θα ήθελα να σας πω το εξής κύριε Ντεβά όμως. Μου είσαστε πολύ συμπαθητικός. Ε, καταρχάς σχετικά με την απεικιοκρατία και μετά με τον πατερναλισμό. Όλες αυτές οι μορφές έχουν αποτύχει, πρέπει να βρούμε νέες διεξόδους και να δεχθούμε τους κινδύνους εφόσον οι προτάσεις υπερβαίνουν τους κινδύνους. Δεν μπορούμε δηλαδή να κάνουμε τίποτα αν δεν αναλάβουμε κάποιον κίνδυνο. Αν είμαστε υπολογιστέ, δεν θα πετύχουμε τίποτα. Με κάποιο καλύτερο συνδυασμό θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Εξού και πιστεύω ότι η δημοσιονομική ε, στήριξη δεν είναι μία επιταγή εν λευκό, είναι ένα μέσο για εξυπηρέτηση ε, της ε, ενδογενούς πολιτικής των κρατών που αποδέχονται τη στήριξη αυτή. Αυτά που είπε ο κύριος Τυρολιά συμφωνώ απολύτως, διότι δεν νομίζω κατά ότι υπάρχει συσχετισμός μεταξύ της αυξήσεως των των ε, ε, χωρών, των, ε, της στήριξης μιας χώρας και της αυξήσεως των στρατιωτικών δαπανών. Βλέπουμε τώρα ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν ενδοεθνικές σειράξεις και ουσιαστικά η αστυνομία χρειάζεται περισσότερη βοήθεια για να λύσει τα προβλήματά της. Επιπλέον βλέπουμε ότι υπάρχει μία περιφερειακή ολοκλήρωση στην Αφρική και ε, υπάρχει μια θεσμική αλλαγή ε, καταρχήν ε, παγκοσμίως με την Αφρικανική Ένωση η οποία αυτή τη στιγμή συμμετέχει στη διαχείριση ασφαλείας διεθνώς και σε το Ευρωπαϊκό ε, Ταμείο Ανάπτυξης που συγχρηματοδοτεί και μετά υπάρχουν ε, οι διάφορες αποφάσεις σχετικά με την ανάπτυξη που απορρέουν από την ασφάλεια και πρέπει αυτή τη στιγμή να λάβουμε υπόψη όλα αυτά τα θέματα και άρα ε, θα πρέπει κάπως ε, να αναθεωρήσουμε τις απόψεις μας ή να ε, ξαναξετάσουμε το θέμα μετά από λίγα χρόνια. Ο, πολύ σωστά μας μιλάει ο κύριος Τυρολιά για αποκέντρωση. Αν όντω υπάρχει ένα μέσον αποκέντρωσης, διότι στην αρχή τα κράτη-μέλη έδιναν λίγα χρήματα στους στοχούς. Στη συνέχεια ε, χρειάστηκε ένας ε, Ολλανδός σοσιαλιστής τον οποίο θαυμάζω πάρα πολύ γιατί οι σοσιαλιστές ήταν πάντοτε ευγενείς μαζί μου κυρία Πρόεδρε και νομίζω ότι στο τέλος ε, της συνεδρίασης θα ζητήσω να τοποθετηθώ προσωρινά δίπλα σοσιαλιστές διότι πρόκειται για μια διαδικασία βαθμιαία. Ε, κάποια στιγμή ελέγχθη ότι δεν θα λύνονται όλα στη Χάγη, αλλά θα αναθέσουμε και εξουσίες εις τις χώρες αποδέκτες της βοηθείας, δηλαδή υπάρχει μια σημαντική αποκέντρωση από τις πρωτεύουσες που εκταμιεύουν προς τις περιοχές που πρέπει να αναπτυχθούν ενδογενώς. Και όπως είπατε κύριε Τυρολιά, δεν αναφερθήκατε εις ε, τις ε, αρχές στις οποίες βασίζω αυτό το σκεπτικό και ε, ελπίζω ότι θα αποδεχθείτε τις απόψεις μου και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία χρησιμοποιεί καινοτόζου μεθόδους στο θέμα αυτό ε, πρέπει να χαιρετιστεί και ε, θα μπορέσουμε για το μέλλον να κερδίσουμε αυτές ε, τις προκλήσεις οι οποίες ε, να αντιμετωπίσουμε οι προκλήσεις που υπάρχουν. 12 Απριλίου το μεσημέρι τελειώνει η προθεσμία των τροπολογιών και περνάμε τώρα εις το σημείο 12 όπου περιμένουν την κυρία Φραντσέσκα Μπαλτσάνη που δεν έχει έρθει και θα επανέλθουμε και στο σημείο 9 Έχουμε 39 ε, τροπολογίες στην έκθεση της κυρίας Κρέζε, εξωτερική διάσταση της κοινωνικής πολιτικής, της πρόθεσης εργασιακών και κοινωνικών προτύπων και κοινωνική ευθύνη των ε, ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Η κυρία Γκρέση ζήτησε ε, να υπάρξει μια ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις τροπολογίες διότι 26 ε, ε, Ιανουαρίου είχε αποφασιστεί από τους συντονιστές ότι οι τροπολογίες θα πρέπει, οι συμβιβαστικές τροπολογίες θα πρέπει να είναι στη γραμματεία στις 13.00 της ε, παραμονής της ε, ε, ε, της ψηφοφορίας. Και άρα τώρα πλέον ό,τι και να πει η κυρία Γκρέσ δεν μπορεί να υπάρξουν ούτε τροπολογίες ούτε αίτηση να ψηφίσουμε χωριστά μία, σε δύο μέρη μία τροπολογία. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αντιλαμβάνομαι ότι δεν υπάρχει ε, πλέον δυνατότητα ε, ελιγμών αλλά νομίζω ότι σκόπιμο θα ήταν να ξανασυζητήσουμε το θέμα. Διότι η βασική ιδέα αυτής, ε, αυτού του θέματος είναι να αλλάξουμε την μεταβλητή γεωμετρία την οποία έχουμε στο θέμα της κοινωνίας και της εργασίας διότι στις ε, ε, κοινωνικές συμφωνίες, πότε μιλάμε για κοινωνικά δικαιώματα, πότε για κοινωνική νομοθεσία και αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι ποτέ δεν μιλάμε για την ε, συνθήκη του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας στις οποίες βασίζονται. Άρα πρέπει να συμφωνήσουμε ότι δεν εφαρμόζεται επαρκώς και τονίζω τον, τον όρο εφαρμογή ε, των κοινωνικών προτύπων, πράγματα το οποίο ε, ε, προσωπεύει μία παγκόσμια άποψη για την, για την, την επίτευξη των στόχων αναπτύξης σε Επίσης υπάρχει η κοινωνική διάσταση σχετικά με την εξωτερική δράση. Ήδη καταφέραμε ε, να διατυπώσουμε πολλές συμβιβαστικές τροπολογίες, αλλά θα ήθελα εδώ να σας πω ότι ορισμένες υποκινήσεις δεν επαρκούν και θα πρέπει να προχωρήσουμε σε μηχανισμούς ε, υποχρεωτικούς και ε, σε νομικές ε, διατυπώσεις. Όλοι γνωρίζουμε τη θεωρία αλλά δεν έχουμε κάποιο μηχανισμό εφαρμοστικό, ενιαία εφαρμοστικά για αυτά τα κοινωνικά πρότυπα. Άρα εδώ διακυδεύεται η αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Αυτά μόνο είχα να σας πω σήμερα το πρωί και σας ευχαριστώ που μου δώσετε το λόγο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ε, εισηγήτρια για την εξαιρετική δουλειά που έκανε. Στα πλαίσια αυτών που έχουμε συζητήσει και στα πλαίσια των νέων τροπολογιών, οι σοσιαλιστές και οι δημοκράτες θέλουν να επιστήσουν την προσοχή ε, σε, ε, στα εξή σημεία. Πρώτον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να προχωρήσει στην διατύπωση μιας κοινωνικής ρήτρας ε, σταθερής, η οποία θα περιλαμβάνεται σε όλες τις συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών που θα συνάπτει και διμερών και πολυμερών. Είναι λοιπόν προς την κατεύθυνση αυτή απαραίτητο οι συμφωνίες που είναι σε στάδιο διαπραγμάτευσης από την Επιτροπή να περιλαμβάνουν αυτές τις κοινωνικές ρήτρε, έτσι ώστε η συμπερίληψη των χωρών αυτών ε, στην ε, διεθνή αγορά να μην γίνεται συστηματικά εις βάρος των εργαζομένων. Ταυτόχρονα η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί έτσι ώστε οι διεθνείς χρηματοδοτικοί μηχανισμοί και οι διεθνείς οργανώσεις να είναι πρότυποι κοινωνικής ευθύνης όταν παραμβαίνουν στις χώρες ε, υποανάπτυξη σχετικά μάλιστα με την παιδική εργασία. Νομίζω ότι είναι απαραίτητο επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συμπεριλάβει περισσότερο τα συνδικάτα και τις ΜΚΟ στις ε, προτάσεις τις οποίες κάνει για την κοινωνική υπευθυνοποίηση των επιχειρήσεων και στον τομέα της εμπορικής πολιτικής, στον ΠΟΕ και στα υπόλοιπα θεσμικά όργανα όπως επίσης και στα προγράμματα τα οποία προέρχονται από τις περιφερειακές συμφωνίες τις οποίες συνάπτει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Το σχέδιο ψηφίσματος θα το ψηφίσουμε στις 3 το μεσημέρι. Περνάμε λοιπόν στο σημείο 8. Εντολή για τριμερή διάλογο για το σχέδιο προϋπολογισμού του 12. Η Επιτροπή Προϋπολογισμών θα ψηφίσει τον Μάιο μια έκθεση η οποία θα καθορίσει τις θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο στα πλαίσια του τριμερούς δημοσιονομικού διαλόγου. Θα πρέπει να δώσουμε τη γνωμοδότησή μας στην Επιτροπή Προϋπολογισμών το μήνα Μάιο για να ακουστούν οι απόψεις ε, ε, των υπολείπων κοινοβουλευτικών επιτροπών εκ των προτέρων. Η κυρία Μπαλτσάνη είναι παρούσα σήμερα εδώ για να ακούσει αυτά τα οποία θα υποθούν και της δίνω το λόγο αμέσως αφού την καλωσορίσω. Σας ευχαριστώ για τη συνάντηση αυτή. Η επεξεργασία του προπολογισμού βρίσκεται στην πρώτη της φάση, μια ευαίσθητη φάση, στα πλαίσια της οποίας επιβάλλεται να προχωρήσουμε και ταυτόχρονα συλλέγουμε ουσιαστικά την πρώτη ύλη που θα μας οδηγήσει στην δυνατότητα απόφασης μιας ε, συνεκτικής και ξεκάθαρης πολιτικής δράσης. Καθορίζονται δηλαδή οι προτεραιότητες του προϋπολογισμού. Φέτος η πρότασή μου, την έχετε δει στο έγγραφο εργασίας ε, που επεξεργαστήκαμε στα μέσα Φεβρουαρίου και το ψήφισμα που θα σας δώσουμε αύριο, προσπαθούμε να διασφαλίσουμε μια κάποια συνοχή στις προτεραιότητες ανάμεσα στις προβλέψεις μας στις δημοσιονομικές για το 12 με τους μεγάλους στόχους που έχουμε για τη στρατηγική του 20. Για τη στρατηγική του 2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει κάποιες συγκεκριμένες μεθοδολογικές επιλογές. Προσπαθεί να συγκεντρώσει την προσοχή και τις δυνάμεις της σε μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη φάση και να εμπλέξει σε εισαγωγικά τα κράτη-μέλη έτσι ώστε να αναλάβουν τις υποχρεώσεις τους σε συγκεκριμένους στόχους. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν ποιοι είναι αυτοί οι κοινοί στόχοι των ευρωπαϊκών χωρών. Στα πλαίσια αυτή τη συγκεκριμένη πλατφόρμας λοιπόν θα πρέπει να βρούμε κάθε χρήσιμο μέσο το οποίο να μας βοηθήσει να βγούμε από μια περίοδο κρίσης ε, στην οποία ζούμε και θα πρέπει ο καθένας στα πλαίσια των δικών του αρμοδιοτήτων να αναλάβει κάποιες, να καθορίσει κάποιες προτεραιότητες, επίγουσες προτεραιότητες που θα πρέπει να διαφαίνονται στον προϋπολογισμό ήδη από το 12. Είναι απαραίτητο λοιπόν και γι' αυτό συνεργαζόμεστα η διαδικασία η δημοσιονομική από την αρχή να βγει από την Επιτροπή Προϋπολογισμού και να καταστεί ένα θέμα το οποίο γίνεται αντικείμενο επεξεργασίας από κοινού από τις εξειδικευμένε επιτροπές, γιατί οι εξειδικευμένε αυτές κοινοβουλευτικέ επιτροπές με τις γνώσεις τους και την αρμοδιότητά τους καθορίζουν, θα έλεγα, το πιο χρήσιμο κομμάτι που θα βοηθήσει στον καθορισμό των προτεραιοτήτων των δημοσιονομικών. Από αυτή τη φάση λοιπόν από τώρα η προσπάθειά μου η δημοσιονομική είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να συζητηθεί σε όλες τις εξειδικευμένες επιτροπές και όλες αυτές να μας βοηθήσουν να καθορίσουμε σωστά ποιες είναι οι πολιτικές, ποιες οι δράσεις και ποια τα προγράμματα τα οποία θα πρέπει να στηρίξουμε με την περισσότερη δύναμη που έχουμε για το 12 στα πλαίσια της στρατηγικής 2020. Ο τίτλος 4 όπου εκεί εντάσσονται τα προγράμματα τα οποία εσάς αφορούν, είναι θα έλεγα αυτή η οποία συστηματικά υποφέρει από υποχρηματοδότηση. Και ακριβώς οι προτεραιότητες τις οποίες έχετε σε σχέση με τις δημοσιονομικές είναι οξύτατες προτεραιότητες, πιστώσεις για να προσδοθεί αξιοπιστία στις δράσεις μας και ταυτόχρονα και η δυνατότητα να υπάρχει μια κάποια ευελιξία έτσι ώστε ο προϋπολογισμός να ανταποκρίνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα στις ανάγκες που υπάρχουν. Γι' αυτό λοιπόν είναι απαραίτητο από τώρα να μπορέσετε να μας υποδείξετε τις προτεραιότητες στα πλαίσια των δικών σας αρμοδιοτήτων και αυτές να εξεταστούν το ταχύτερο δυνατόν. Μέχρι τον επόμενο Ιούνιο, σαν παράδειγμα, τελειώνει η προθεσμία για την προετοιμασία των προπαρασκευαστικών δράσεων είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί αντιπροσωπεύουν θα έλεγα τη δική μας κοινοβουλευτική δυνατότητα πρωτοβουλίας και ταυτόχρονα δίνουν και μια πολιτική θα έλεγα εικόνα στον ίδιο τον προϋπολογισμό. Οι προπαρασκευαστικές αυτές δράσεις είναι αναπόσπαστο τμήμα ε, των δυνατοτήτων τις οποίες έχουμε και είναι ουσιαστικά και το πρώτο πέρασμα μέσα από το οποίο θα προσπαθήσουμε να θέσουμε σε λειτουργία τις προτεραιότητες τις οποίες ακόμα δεν καθορίσαμε. Πρόσκλησή μου λοιπόν είναι να εξετάσετε τα πιλωτικά προγράμματα και τις προπαρασκευαστικές δράσεις έτσι ώστε να δούμε ποια θα πρέπει να υποστηριχθούν και ποια όχι πριν κατατεθούν νέα προγράμματα. Υπάρχει επίσης η προθεσμία της 20 Απριλίου. Μέχρι τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα λάβει υπόψη τις δικές σας δημοσιονομικές προτάσεις και θα επιτρέψει από εκεί και πέρα μια διασταυρούμενη μορφή ανάπτυξης των προτάσεων για τον προϋπολογισμό τους επόμενους μήνες. Σταδιακά, μετά από αυτή τη φάση, μπορούμε να καταθέσουμε τις τροπολογίες μας. Όλα αυτά τα στάδια λοιπόν θα αποδειχθούν πιο αποτελεσματικά εφόσον υπάρχει μια πολιτική σταθερότητα στις απόψεις τις οποίες έχουμε. Σας καλώ λοιπόν να υιοθετήσετε σε εισαγωγικά τον προϋπολογισμό, να τον θεωρήσετε δικό σας και να μας υποδείξετε από τώρα ποιες είναι οι πολιτικές γραμμές και οι συγκεκριμένες θέσεις οι οποίες για σας θέλετε να γίνουν πραγματικότητα για το 12. Γκέρενς έχει το λόγο. Να ευχαριστήσω τη Γενική Συγγήτρια για τον προϋπολογισμό, καθόρισε το γενικό πλαίσιο μέσα στο οποίο καλούμεθα να κινηθούμε. Μας βοηθά να καθορίσουμε τις προτεραιότητες μας στο δημοσιονομικό κομμάτι, στον τομέα της συνεργασίας και για την ανάπτυξη. Θα ήθελα να κάνω δύο τύπου παρατηρήσεις. Οι πρώτες αφορούν τις προτεραιότητες και οι δεύτερες τη μέθοδο. Σχετικά με τις προτεραιότητες μας, αυτές που θα ήθελα να σας υποβάλω, δηλαδή είναι οι εξής. Πρώτον, ότι έχει σχέση με την μετρίαση των κλιματολογικών συνεπειών στις υποανάπτυξη χώρες. Θα πρέπει εκεί να πούμε ότι οι πιστώσεις θα πρέπει να είναι επιπλέον. Αυτή είναι μια παρατήρηση την οποία θα πρέπει να την επαναλαμβάνουμε συνεχώς. Δεν θα πρέπει να κουράζεται κανείς να την ακούει γιατί είναι απαραίτητο να γίνει πραγματικότητα. Και οι εξηγήσει τις οποίες μας έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή νομίζω ίσως να καθησυχάσουν αυτούς οι οποίοι θεωρούν ότι μπορεί να υπάρξει μια σύγχυση ανάμεσα σε δύο διαφορετικούς τομείς. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να δουν το θέμα με τον ίδιο τρόπο και δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση η προτεραιότητά μας αυτή να φυγεί. Γιατί αλλιώς στην περίπτωση την διαφορετική απλά θα υπάρξει μια διαφορετική ονομασία συγκεκριμένων κεφαλαίων και όχι επιπλέον χρήματα. Τώρα για μη συγκεκριμένου όπως τις μπανάνας, εδώ θα πρέπει να μιλήσουμε για επιπλέον πιστώσεις, γιατί αλλιώς για μια ακόμη φορά θα επιβαρύνουμε τα λεγόμενα αναπτυξιακά ε, μέσα συνεργασίας. Είναι μια δυναμική η οποία έχει δημιουργηθεί στις χώρες ΑΚΕ και τώρα οι χώρες ΑΚΕ στερούνται των πλέον εκτιμάτων των, ε, των, ε, των, των εμπορικών προτιμήσεων και των ειδικών καθεστώτων. Τρίτον, θα πρέπει να συγκεντρώσουμε την πολιτική ανάπτυξη για τη συνεργασία στις πιο σημαντικές ανάγκες, στους τομείς που παρουσιάζουν τις πιο σημαντικές ανάγκες. Θυμίζω εδώ τις συζητήσεις τις οποίες είχαμε για το θέμα της εφαρμογής των μέσων ε, συνεργασίας για την ανάπτυξη. Οι χώρες σαν τη Βραζιλία δεν έχουν ανάγκη να δοθούν χρήματα στα πλαίσια αυτά. Η Βραζιλία μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες της για την καταπολέμηση της φτώχειας με τους ίδιους του πόρους. Δεν πρέπει άλλοι να χρηματοδοτήσουν γιατί η οικονομία της Βραζιλίας έχει πόρους και έχει υψηλότατους ρυθμούς ανάπτυξης. Θα πρέπει λοιπόν στο τέλος της διαδικασίας όταν όλα αυτά τα αναπτυξιακά μέσα ε, συνεργασίας ε, ε, ξεδιπλωθούν θα πρέπει να διαλέξουμε να δούμε ποιοι είναι αυτοί που έχουν τις μεγαλύτερες ανάγκες και αυτούς να στηρίξουμε. Τέταρτον, οι συζητήσεις για τις εμπορικές συναλλαγές. Εδώ θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε λίγο. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να θίξουμε τους στόχους το 0,7% σχετικά με το ΑΕΠ, ποσοστό του ΑΕΠ. Αυτός ο στόχος το 0,7 του ΑΕΠ θα πρέπει να παραμείνει ένα στόχος και ένα κεκτημένο της Ένωσης. Οι στόχοι αυτοί θα πρέπει να επιτευχθούν μέχρι το 2015 γιατί αλλιώς στην ουσία προκαλούμε μια ρήξη στην πολιτική μας γραμμή και δεν έχουμε το ηθικό δικαίωμα να το κάνουμε. Μια πέμπτη προτεραιότητα εγγραφόμενη στα πλαίσια της ανθρωπιστικής δράσης και της προστασίας του πολίτη. Η συνθήκη της Λισαβόνας εδώ δίδει νέες δυνατότητες θα πρέπει της πολιτικής προστασίας, συγγνώμη όχι της προστασίας πολίτη. Εδώ θα πρέπει και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε επίπεδο εθνικό να γίνουν συνεργασίες, κάτι το οποίο θα μας επιτρέψει και να εξοικονομήσουμε χρήματα και να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί. Θα πρέπει επίσης να διατηρήσουμε την χρηματοδότηση των διεθνών ταμείων για την καταπολέμηση της ελονοσίας, του AIDS και της φυματίωσης. Νομίζω ότι εδώ κάποιες φορές ακούγονται διστακτικές για τη χρηματοδότηση του Ταμείου για το AIDS, σαν παράδειγμα, γιατί έχουν δημιουργηθεί ορισμένα προβλήματα. Να θυμίσω ότι το ίδιο το Ταμείο έφερε στην επιφάνεια τα προβλήματα αυτά. δεν συλλάβαμε κάποιον επαυτοφόρο, οι ίδιοι ε, ε, εξεπλάγησαν από αυτό που είδαν και το έφεραν στην επιφάνεια. Είναι αποκαλυπτικό της κατάστασης που δημιουργεί, αλλά δεν θα πρέπει αυτό να λειτουργήσει εις βάρος τους. Αυτό θα ήταν ιδιαίτερα άδικο. Επαναλαμβάνω αυτό το οποίο είπα το πρωί. Ε, όλα όσα πράττουμε παρουσιάζουν κινδύνους. Δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση κάτι το οποίο να είναι ε, αμέτωχο κινδύνων. Θα πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε ε, την το ταμείο αυτό για το AIDS, γιατί ακριβώς η αποκάλυψη μιας απάτης εξηγεί και αποδεικνύει ότι υπάρχει ένα σύστημα ελέγχου. Το δεύτερο τμήμα λοιπόν της παρέμβασής μου αφορά τη μέθοδο. Αναφέρθηκε η συγγήτρια στο κεφάλαιο 4. Πιστεύω ότι τα χρήματα τα οποία δεν χρησιμοποιούνται δεν θα πρέπει να επανέρχονται στα κράτη-μέλη, αλλά να συμπληρώνουν επιστώσει, οι οποίες έχουν πάρα πολύ μεγάλες ελλείψεις. Πάντα σε σχέση με τη μέθοδο, οι λεγόμενες διοικητικέ δαπάνε. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι σε θέση να φέρει πέρα στην αποστολή τη, έχοντας πάντα τις απαραίτητες δυνατότητες σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού αυτό ακούγεται ε, λίγο περιττό, αλλά παρόλα αυτά είναι ένα επαναλαμβανόμενο αίτημα, ιδιαίτερα τεκμηριωμένο και θα πρέπει να το παρουσιάσουμε. Θα ήθελα κλείνοντας να πω ότι χάσαμε μια ευκαιρία μέσω της σύμπτυξης της Γενικής Διεύθυνσης Συνεργασίας με το ΕΚΟ. δεν θέλω εγώ να αμφισβητήσω το, το, τη σωστή λογική αυτής της αντίληψης, αλλά νομίζω ότι θα έπρεπε να υπάρξει στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ένας πυρήνας ανεξάρτητος επεξεργασίας θέσεων για την βοήθεια και την ανάπτυξη που θα μπορούσε να εμπλουτιστεί από τη συνεισφορά των υπαρχόντων ίδιων οργανισμών να συνθέσει τις θέσεις αυτές και να εμπλουτίσει με τη σειρά του την πολιτική μας για την ανάπτυξη σαν Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει ανάγκη από επιστημονικά σταθερά θεμέλια. Λοιπόν, αυτά είναι τα εννέα σημεία που ήθελα να θέσω. Τα έξι αφορούν ε, τις προτεραιότητες, τα τρία αφορούν την μέθοδο και ελπίζω να μπορέσουμε έτσι να βοηθήσουμε να τα απορροφήσει η συγγήτριά μας. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Ντέβα, ζητήσετε το λόγο. Να είστε σύντομος, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ σημαντικό που ήρθατε να μας πείτε σε μια πρώιμη φάση, τι είδου ε, καταχρήσεις γίνονται στο προπολογισμό. Και αυτό δείχνει πόσο αξιόπιστη είναι η εργασία που γίνεται εδώ. Αλλά αυτό το οποίο με ανησυχεί είναι ότι καμιά φορά δεν εξετάζουμε αυτό το οποίο πετύχαμε ή δεν επιτύχαμε σε μια περίοδο 10 ετών επί παραδείγματα. Ε, εργαζόμαστε εδώ και 35 χρόνια σε αυτό το τομέα. Και αν δούμε τους τρόπους που σπαταλήθηκαν τα χρόνια στη λεγόμενη ανάπτυξη, διαπιστώνουμε ότι πρόκειται για περίπου 500 δισεκατομμύρια ευρώ που αφορούν την παροχή οικονομικής βοήθειας προς τις φτωχότερες χώρες του κόσμου αλλά σε όλες αυτής της ε, περίοδου ε, τελικά δεν διαπιστώνουμε ότι πραγματικά με τα χρήματα αυτά εξαλείψαμε τη φτώχεια. Και ίσως ε, δεν επικεντρώσαμε, δεν συστήκαμε σε άλλες χώρες, όπως είναι για παράδειγμα το Βιετνάμ, η Ταϊλάνδη, η Ινδονησία και η Κίνα η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν βοήθησε αυτές τις χώρες την εξάλληψη της φτώχειας γιατί δεν επικεντρώσαμε τις προσπάθειες τόσο όσο στην Αφρική, την Καραϊβική, τις χώρες του Ελληνικού ή άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής. 380 δισεκατομμύρια άνθρωποι ε, ζουν στις φτώχεια στην Κίνα, το Βιετνάμ, την Ινδονησία κλπ. Και υπάρχει μια μείωση του ΑΕΠ σε έξι χρόνια, μαχτική μείωση. Νομίζω ότι δεν ε, προβληματιζόμαστε αρκετά για το τι γίνεται όσον αφορά την εξέλιξη φτώχεια. Τι κάνουν ορισμένε χώρε που τελικά βγαίνουν από τη φτώχεια, ενώ άλλε παραμένουν καθυλωμένε, τελματώνονται μέσα στην ε, φτώχεια. Ε, νομίζω ότι ε, θα πρέπει να έχουμε μια μακροπρόθεσμη ανάλυση των προσπαθειών μας ε, για να μην συνεχίσουμε να κάνουμε το ίδιο τα επόμενα χρόνια. Ίσως θα μπορούσαμε να προβληματιστούμε σε σχέση με τον αντίκτυπο που έχουν οι προσπάθειές μας ή την έλλειψη ακριβώς αντικτύπου. Ε, κάποιες χώρες πραγματικά έγιναν πιο πλούσιες χωρίς τη βοήθειά μας. Το λόγο έχει η Επιτροπή, ο κύριος Μάρτιν Πέμιγκτον. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομος. Χαιρετίζουμε τη συζήτηση αυτή και λαμβάνουμε γνώση ε, των ανησυχιών της Επιτροπής και αναμένουμε ανυπομονησία την ανάπτυξη μιας καλής ε, συνεργασίας με τον εισηγήζο ότι αυτή ήταν από τις πιο πετυχημένες ε, θητείες της Επιτροπής αυτής όπου μπορέσαμε πραγματικά να συζητήσουμε ε, για θέματα που μας ανησυχούν από κοινού. Η Επιτροπή βρίσκεται στη φάση οριστικοποίησης του σχεδίου προπολογισμού που θα είναι έτοιμο σε ένα μήνα. Και ε, νομίζω ότι μέχρι τότε μπορούμε να κανονίσουμε κάποιες συναντήσεις για να συζητήσουμε λεπτομεριακά κάποια επιμέρους θέματα. Σας ευχαριστώ, εν πάση περιπτώσει, για τις εισφορές σας που υπήρξαν ιδιαίτερους πολύτιμες. Η κυρία, η θέλετε να πάρετε το λόγο για να ολοκληρώσετε. Σας ευχαριστώ λοιπόν για τις πολύ σημαντικές σας ιδέες, αν και όλες πολύ στενά συνδεδεμένες με το θέμα μας. Αναφέρθηκα και στο θέμα της καταπολέμησης των συνεπειών των κλιματολογικών αλλαγών, καταπολέμησης των ασθενειών, καταπολέμησης της ένδυας και τέθηκε κι άλλο ένα θέμα σημαντικό, η ανάγκη η οποία υπάρχει να υπάρξουν επιπλέον πόροι, κάτι το οποίο δεν το λέμε συχνά ή να μην χρησιμοποιούνται σαν παράδειγμα οι επιστροφές και τα μη χρησιμοποιηθέντα ποσά και πιστώσεις. Όλα αυτά είναι κάτι που λειτουργούν αρνητικά στις πολιτικές μας, ιδιαίτερα όταν δεν ενισχύουμε τις υπόλοιπες πολιτικές. Αναφέρθηκε επίσης και η ανάγκη επαναδιατύπωσης των προτεραιοτήτων ε, που θα καθορίσουν τις πολιτικές μας. Όλα αυτά τα θέματα είναι κεντρικά για τον προϋπολογισμό και είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να συγκεκρινοποιήσω κατά τη διάρκεια της δημοσιονομικής διαδικασίας, Μια διαδικασία που όπως είπα στην αρχή της παρέμβασής μου θα πρέπει να, να, εξαχθεί, να διεξαχθεί θα έλεγα σε πάρα πολύ στενή και γειτονική σχέση ανάμεσα στην Επιτροπή Προϋπολογισμών και τις εξειδικευμένες λεγόμενες επιτροπές. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Γκέρνς έχει το λόγο. Και εγώ ίδιο θα ήθελα να επισημάνω ένα στοιχείο. Ο κύριος Ντέβα επέμεινε επίση την ανάγκη ε, να προβληματιστούμε ε, σε σχέση με την ε, πολιτική ανάπτυξη και των πραγματικά μέτρων αποτελεσμάτων παρήχθησαν σε ορισμένε χώρε. θα ήθελα να φέρω κάποιου αριθμού, νομίζω ότι ήδη το έπραξα το 81 μέχρι το 2011 υπάρχει μια ανάπτυξη του παγκόσμιου ΑΕΠ περίπου 19 δισεκατομμύρια δολάρια και σύμφωνα με μια έρευνα μόνο 2% αυτού του ποσού δημιουργίας νέου πλούτου τελικά έληξε στους πιο φτωχούς. Αλλιώς δεν θα είχαμε όλους τους φτωχούς που ζούμε κάτω από 2 δολάρια τη μέρα. Παραδέχομαι ότι δεν μπορούμε να επιλύσουμε το πρόβλημα αυτό μόνο με τα μέσα του προπολογισμού, με δημοσιονομικά μέσα, αλλά πραγματικά αφορά τη συνεκτικότητα των πολιτικών μας. Για παράδειγμα, έκθεση Ζολή, ε, στα τελευταία ολομέλεια. Οι χρηματοοικονομικές ροές, το φαινόμενο διαφθοράς, ε, το ζήτημα που τέθηκε εδώ, η θεσμική ικανότητα αυτών των χωρών όλοι αυτοί οι παράγοντες. Και για να σας ε, καθησυχάσω όσον αφορά την προσέγγιση αυτών των θεμάτων. Ίσως είναι κάτι το οποίο απλώς ονειρεύουμε, ένα όραμα που έχουμε. Ίσως οι επιστημονικές έρευνες μπορέσουν να μας επιτρέψουν μια βελτίωση. Καμιά φορά υπάρχουν κάποιες διχογνωμίες όσον αφορά τα βασικά στοιχεία τα οποία θα πρέπει να έχουμε στη διάθεσή μας δεν είναι αυτή η μόνη επιτυχία, αλλά νομίζω θα πρέπει να μείνουμε εδώ και θα πρέπει να δείξουμε κάποια υπομονή. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και θα ήθελα να ρωτήσω την Επιτροπή εάν μπορώ να συνεχίσω να εργάζομαι πάνω στις προτεραιότητες που διατύπωσα και στα τρία, τις, τρεις, ε, τα τρία σημεία της μεθοδολογίας ε, δεν θα ήθελα... Ε, θα πρέπει η Επιτροπή να αποδεχτεί αυτές τις ε, προτεραιότητες και δεν ξέρω κατά πόσο είμαστε σε θέση να ισχυριστούμε κάτι τέτοιο. Ε, ευχαριστούμε πολύ. Θα περάσουμε τώρα στο τελευταίο σημείο της ημερήσιας διάταξης, το σημείο 10 τη μελλοντική συνεργασία μεταξύ τοπικών αρχών και μη κρατικών φορέων. Ε, αφορούν ε, τη συζήτηση για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας στα θέματα αυτά. Α, και έχουν σαν σκοπό να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα του, του συνόλου των ε, δρόντων στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας. Η αποτελεσματικότητα της ε, διεθνούς ε, βοήθειας δίδεται στην κοινωνία των πολιτών και στις τοπικές αρχές ένα καινούριο ρόλο που δεν περιορίζεται στην εφαρμογή των προγραμμάτων αλλά περιλαμβάνει επίσης την συμμετοχή στη διατύπωση των πολιτικών ανάπτυξη. Υπό την έννοια αυτή η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και των τοπικών αρχών συνιστά ένα σημαντικό βήμα προς τα Προ προς την πορεία του εκδημοκρατισμού και της αυτοδιάθεσης. Η δήλωση των Παρισίων προβλέπει ε, την ευθυγράμμιση των πολιτικών των δωρητριών χωρών στις πολιτικές των χωρών ε, εταίρων που αποδέχονται τη βοήθεια. Οι πολιτικές αυτές θα πρέπει να καταρτιστούν μέσω μιας δημοκρατικής διαδικασίας που περιλαμβάνει την κοινωνία των πολιτών η έννοια του ownership είναι κάτι παραπάνω από μια οικειοποίηση αυτή της δυνατότητας του δυναμικού εκ μέρους των ε, χωρών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή που ξεκίνησε αυτή τη διαδικασία, η οποία συνενώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τι χώρε μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώ και τι οργανώσει τη κοινωνία των πολιτών και τι τοπικέ αρχέ, καθώ και αυτέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο αυτέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και των χωρών εταίρων μα. Ο κύριο ε, Μπάλιο της Γενικής Διεύθυνσης ΤΕΦΚΟ της Επιτροπής θα μας ε, παρουσιάσει τα αποτελέσματα αυτής της μακράς διαδικασίας διαβούλευσης και των μελλοντικών της προοπτικών. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στον κύριο Μπάλιο. Yes, Καλημέρα σας ε, όλοι. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές, Επιτρέψατε μου καταρχήν να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την υποστήριξη που παρέχει σε αυτή τη ε, διαδικασία και για την συμμετοχή ορισμένων μελών του Κοινοβουλίου σε, αυτή, σε αυτό το δύσκολο έργο των ε, ομάδων εργασίας και των περιφερειακών ε, σεμιναρίων. η συμμετοχή αυτή προσλαμβάνει ιδιαίτερα δυναμικό χαρακτήρα και εμπλουτίζει πραγματικά την ποιότητα της ε, συζήτησης. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Πρόεδρο ε, ε, για την πρόσκληση των μάδων εργασίας τον Ιανουάριο, όπου θεωρώ ότι ο διάλογος ήταν ιδιαίτερα σημαντικός. Όπως υπενθυμίσατε ήδη, κυρία Πρόεδρε, ο διαρθωμένος ε, διάλογος είναι μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε από τον Επίτροπο κύριο Πίλμπαξ τον ε, περασμένο Μάρτιο του 2010 για να συζητήσει συμπερίληψη των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των τοπικών αρχών στην αναπτυξιακή πολιτική. Αυτό γίνεται σε μια μόνιμη βάση και επίση συμμετέχει το Συμβούλιο στι συζητήσεις αυτέ ορισμένε φορέ, Πρόκειται για μια εις βάθος και πολύ τεχνική προσέγγιση. Θα ήθελα επίσης να σε επενθυμίσω ότι το ζήτημα των μη κρατικών φορέων και των τοπικών αρχών στην ε, στο επίπεδο της ανάπτυξης, στον πέρα της ανάπτυξης της συνεργασίας δεν αφορά μόνο τον τρόπο χρηματοδότηση των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Το ζήτημα, τα ζητήματα είναι πολύ πιο σημαντικά και πλατιά κατά την άποψή μας. Και τα τελευταία συμβάντα στην Βόρεια Αφρική και στη Μέση Ανατολή μας υπενθυμίζουν αυτό το γεγονός. Ε, δεν είναι δυνατόν να υπάρξει ανάπτυξη χωρίς τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και των ενώσεων της. Αυτή είναι μια πραγματικότητα τόσο στην Ευρώπη όσο και σε όλες τις άλλες περιοχές του κόσμου. Και ορισμένες φορές ε, ε, ίσως να λησμονούμε αυτές τις βασικές αρχές. Η συζήτηση ξεκίνησε προκειμένου να δημιουργηθεί ένας χώρος διαλόγου. Στις Βρυξέλλες αλλά και επίσης σε περιφερειακό επίπεδο. Και αυτό και ακολούθησαν ε, ορισμένες εκθέσεις για τους τρόπους χρηματοδότησης, για παράδειγμα εκ μέρους του ελεγκτικού συνεδρίου ή επίσης τη συζήτηση για την απαλλαγή του 2008, αλλά και τη συστάσεις του Συμβουλίου για την απαλλαγή του 2008. Το ζήτημα και βασική ιδέα ήταν πραγματικά να συσταθεί μια δυνατότητα ε, διαβούλεσης και διαλόγου ακόμα και σε τεχνικά θέματα. Και έγιναν μέχρι στιγμής 6 συνεδράσεις στις Βρυξέλλες και 7 περιφερειακά σεμινάρια στην Αφρική, στη Λατινική Αμερική, την Ασία ε, και την ε, και ε, ε, ε, ε, πραγματικά υπήρξε ευκαιρία να σε τι βάθος το ζήτημα της ανάπτυξης, της εκπαίδευσης και της αύξησης της ειδοποίησης στην Ευρώπη, προκειμένου να προεχθεί και να υποστηριχθεί η έννοια μιας παγκόσμιας θαγένειας. Και τον Ιούλιο 2010 έγινε ένα σεμινάριο τριών ημερών σε σχέση με θέματα που συνδέονται με ζητήματα εκδημοκρατισμού ε, και το, του ρόλου των μη κυβερνητικών οργανώσεων και της κοινωνίας των πολιτών. Επίσης όσον αφορά το ρόλο των τοπικών αρχών στην αναπτυξιακή διαδικασία ε, ε, οι αρχές αυτές βρίσκονται πολύ κοντά ε, στον πολίτη και σε ένα επίπεδο όπου είναι πραγματικά σε θέση να δουν τις ε, ανάγκες των πολιτών. Έχουμε συστήσει τρεις ομάδες εργασίας ε, και αυτός ήταν ένας μόνιμος τρόπος εργασίας μέχρι στιγμής. Η ομάδα εργασίας υπαριθμών 1 που εξετάζει το ρόλο και την προσθέμενη αξία των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και τοπικών αρχών, μια ομάδα η οποία συστάει τη συμπληρωματικότητα και την ε, συνεκτικότητα με τους στόχους της ε, αναπτυξιακής ατζέντα και τα συμπεράσματα αυτών των δύο ομάδων εργασίας ε, αξιοποιήθηκαν για να τροφοδοτήσουμε τη συζήτηση για τον μηχανισμό παροχής βοήθειας που ήταν περισσότερο μια συζήτηση τεχνικής ε, φύσεως αλλά βασιζόμενη ακριβώς στις ε, ανάγκες που εκφράζονται από τις ε, οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών. Για να απαντήσω στην παράκληση του κ. Γκέρνς να είμαστε πιο ταπεινόφρονες ε, θα ήθελα να αναφερθώ στη μεθοδολογία και την προσέγγιση που ακολουθούμε. Πιστεύουμε ότι δημιουργήσαμε μια πολύ θετική δυναμική ε, τάση και είχαμε ανοιχτέ συζητήσεις σε σχέση με το ρόλο τοπικών αρχών ε, και των φορέων αυτών. Σήμερα μπορούμε να κρίνουμε ότι πάνω από 800 συμμετέχοντες με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο συνεισέφεραν ε, στις συζητήσεις αυτές. Η συζήτηση αυτή καθ' αυτή ε, ήταν ιδιαίτερως αξιόλογη και όλες οι εκθέσεις σχολιάστηκαν και αξιολογήθηκαν από όλους τους ε, συμμετέχοντες. Νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι κατά πάσα πιθανότητα αυτή είναι η πρώτη φορά όπου η Επιτροπή και όλοι οι άλλοι ενεχόμενοι υποστηριζόμενοι από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεσμεύονται σε, ένα, σε μια συζήτηση τόσο ανοιχτή και που πηγαίνει εις με την κοινωνία των πολιτών και τις τοπικές αρχές. Δεν πρόκειται για ένα φόρουμ διαπραγμάτευσης εδώ, αλλά όλες οι επιπτώσεις της συζήτησης αυτής αυτού του διαλόγου βεβαίως θα έχουν μείζονες επιπτώσεις κατά την άποψή μας για τις ε, μελλοντικές μορφές συνεργασίας με τις τοπικές αρχές και την κοινωνία των πολιτών συμπεριλαμβάνοντας ελπίζουμε όταν ε, συζητούμε για το πολιετές ε, χρηματοπιστωτικό πλαίσιο τα θέματα αυτά. Τώρα, τι διδάγματα αντλήσαμε. Εάν θέλουμε να αναφερθούμε στη συζήτηση και τα συμπεράσματα της ομάδας εργασίας υπαρχών 1, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει ξεκάθαρα η ανάγκη ενίσχυσης του πολιτικού διαλόγου. Και αυτό είναι αναγκαίο προκειμένου να υπάρξει ένας διάλογος μεταξύ χωρών ε, μελών αυτών των οργανώσεων αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, γιατί οι φορείς ε, της κοινωνίας των πολιτών θέλουν να ενισχυθεί ο πολιτικός τους ρόλος Ταυτόχρονα η οργανώση των κοινωνία, της κοινωνίας των πολιτών και των τοπικών αρχών θα πρέπει να προβούν σε μία αυτοκριτική προκειμένου να βελτιώσουν τους μηχανισμούς αυτοδιαχείρισης που να επιτρέπει μία δυνατότητα λογοδοσίας ε, και διαφάνειας ε, κυρίως ε, στη σχέση με τους χορηγούς και τους δωρητές. Το ίδιο ισχύει και για τις τοπικές αρχές Και πραγματικά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ανοιχτόμυαλη ε, προσέγγιση. Οι ευρωπαϊκές τοπικές αρχές θα πρέπει να δούνε ποια είναι η προστιθέμενη αξία σε αυτές τις εταιρικές σχέσεις, αλλά επίσης να προσπαθήσουν να αποφύγουν τον ανταγωνισμό με τις τοπικές αρχές της, ε, ε, της κοινωνίας των πολιτών Ξέρετε ότι υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους οι ευρωπαϊκοί μη κυβερνητικοί οργανισμοί είναι αυτοί οι οποίοι προσελκύουν τα περισσότερα κονδύλια. σε σχέση για παράδειγμα με το πρόγραμμα για τους μη κρατικούς ε, φορείς. Ταυτόχρονα θα πρέπει να ληφθεί περισσότερο, να ληφθεί περισσότερο υπόψη οι προτεραιότητες των ε, διαφόρων ε, τοπικών ε, φορέων και της κοινωνίας των πολιτών ιδιαίτερα όταν το ζητούμενο είναι να ενισχυθεί μακροπρόθεσμα η η συνεργασία όσον αφορά την ομάδα εργασίας 2 ε, προκειμένου να γίνει μια ανάλυση της ε, συμβολής τους για πιο αποτελεσματική ανάπτυξη ε, θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην ανάγκη διαφύλαξης μιας δυνατότητας δράσης με έναν ανεξάρτητο τρόπο. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα θα κάνουμε υπέρ της ε, κοινωνίας των πολιτών. Και με αυτόν τον ανεξάρτητο τρόπο θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε και πρέπει να το σεβαστούμε ακόμη και αν δεν συνάδει με τις κυβερνητικές προτεραιότητες για να ενισχύσει κανείς τις δυνατότητες μιας χώρας κατά τρόπον ώστε να μπορέσει να έχει τη διαπραγματευτική ε, θέση και την ε, ικανότητα να διαπραγματευτεί με ε, τους δωρητές σε διάφορα επίπεδα. Αυτό αναφέρεται στην διακήρυξη των Παρισίων και το οποίο δεν μπορεί να αντιμετωπίσει κανείς σφαιρικά, πρέπει να το προσαρμόσει σε κάθε περιφέρεια. Και γι' αυτό θέλω εδώ να το συνδυάσω με τον τοπικό παράγοντα διότι αυτό που έχει σημασία είναι ο καθένας να μπορέσει να επέμβει σε τοπικό επίπεδο και ε, να αντιταχθεί στο πρόγραμμα διακυβερνήσεως. Θα πρέπει συγχρόνως να αναπτύξουμε διάφορους επιλεκτικούς μηχανισμούς κατά τρόπον ώστε να ανταποκριθούμε πιο αποτελεσματικά στις ανάγκες οργανώσεως της κοινωνίας των πολιτών ε, όσον αφορά τα επόμενα βήματα θα ξεκινήσουν την επόμενη εβδομάδα με συμμετοχή ορισμένων μελών αυτής της Επιτροπής και θα ολοκληρώσουμε ε, το τέλος Μαρτίου το οποίο έχουμε συνδυάσει με την ε, οργανωμένη συνεργασία κατά τρόπον ώστε να καταλήξουμε στα σωστά αποτελέσματα. Ελπίζουμε ότι στη Βουδαπέστη, στο τελικό σεμινάριο που θα οργανωθεί 17-19 Μαΐου, θα μπορέσουμε να ε, συζητήσουμε με όλους τους εμπλεκόμενους ενδιαφερόμενους για να διατυπώσουμε μία τελική διακήρυξη. Ελπίζουμε να ε, είναι πολιτικές ε, παρατηρήσεις, ε, δεν θα είναι βέβαια δεσμευτικές, αλλά θα είναι σημαντικές και για το μέλλον Εξού και θα θέλαμε, ε, ε, εφόσον μπορεί το Κοινοβούλιο, να προσυπογράψει αυτή την κοινή διακήρυξη στο τέλος του σεμιναρίου της Βουδαπέστη, που δεν θα είναι το τέλος της ιστορίας, αλλά το κλείσιμο μίας φάσεως και άνοιγμα μίας νέας φάσης συνεργασίας με την κοινωνία των πολιτών και τις τοπικές αρχές. Ευχαριστώ. Ο κύριος Νόησεν έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα... Δεν θέλω να προσθέσω κάτι ως προς το περιεχόμενο, γιατί η Επιτροπή μας τα είπε όλα. Σκέφτομαι όμως ότι επειδή έχω συμμετάσχει σε διάφορα περιφερειακά σεμινάρια, ότι ε, θα μπορούσα να εκφράσω αυτό το πνεύμα της συνάντησης διότι ε, δεν είχε μόνο σημασία τι έγινε αλλά ποιος ήταν και πριν και τι έγινε μετά. Δηλαδή υπήρχε μία διασύνδεση μεταξύ των συμμετεχόντων στην κοινωνία των πολιτών και αυτό είναι πολύ σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στην τελευταία περιφερειακή ε, συνάντηση ήταν η εποχή όπου έπεσε, άλλαξε η κατάσταση στην Αίγυπτο. Θελήσαμε να βοηθήσουμε την κοινωνία των πολιτών και θέλω γι' αυτό να ευχαριστήσω τον κύριο Μπάλιο, όχι γιατί κάθε δίπλα μου, αλλά γιατί πρόθυσε το διάλογο αυτό πάρα πολύ. Επίσης και η ομάδα του και προώθησε τις συζητήσεις ε, και με τις γυναίκες και πιστεύω ότι προχωρήσαμε πολύ στη συνεργασία μας και θα αποδειχθεί αυτό και στο επόμενο σεμινάριο της Βουδαπέστης. Ο κύριος Ντέβα έχει το λόγο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω λοιπόν τον εισηγητή για την παρουσίασή του. Πράγματι δείξατε ότι έχετε μπλακεί πλήρω τη διαδικασία αυτή και την κάνετε επίσης και πιο διαφανή για μας. Μία απλή ερώτηση. Η αντιμετώπιση της φτώχειας περνάει από την δημιουργία πλούτου από παράγοντες που γνωρίζουν πώς να δημιουργούν τον πλούτο και μπορούν να τον διανύμουν. Ε, στις ε, προσπάθειες ορισμού που κάνετε για την κοινωνία των πολιτών ε, περιέχετε επίσης και τον επιχειρηματικό κόσμο, τους δημιουργούς επιχειρήσεων, αυτούς οι οποίοι διευκολύνουν γενικά την δημιουργία πλούτου και που ξέρουν ακριβώς ε, να κρατούν βιβλία, ε, να κατανοούν την αξία τους, ε, να κατανοούν την σωστή προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων. Όλα αυτά είναι τμήματα της προσπάθειας δημιουργίας πλούτου. Λοιπόν, χρησιμοποιείτε λοιπόν αυτή την κατηγορία παραγόντων στον μηχανισμό που προβλέπεται για την αντιμετώπιση της φτώχειας. Κύριε Κέλλα. Και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρωτοβουλία της. Είναι πολύ χρήσιμη και περιμένω να δω ποια θα είναι τα αποτελέσματα τα οποία θα χρησιμοποιούμε και εμείς. Συμφωνώ μαζί σας ότι αυτό δεν είναι παρά μόνο το πρώτο βήμα και θα πρέπει να ξεκινήσει μια νέα εποχή η οποία να βασίζεται στα μαθήματα του διαφρομένου διαλόγου και να τα εξελίξει. Θα ήθελα να μάθω αν έχετε συγκεκριμένες ιδέες για τον τρόπο που θα συνεχίσουμε από εδώ και πέρα. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να συζητάμε όταν έχουμε μπροστά μας τον προϋπολογισμό του 2012 ή το πολιετές πλαίσιο. Έχει σημασία αυτό ακόμα και για τον καθορισμό των αριθμών. Έχετε λοιπόν κάποιες συγκεκριμένες ιδέες για το πώς θα εφαρμοστούν όλα αυτά και πώς θα βελτιωθεί η κατάσταση. Ο κύριος Λάστρα. Ε, κύριε Πρόεδρε, καταρχήν θα ήθελα να συγχαρώ την Επιτροπή για την πραγματικά σημαντική εργασία. Θα ήθελα επίσης να σας κάνω μία ερώτηση σε σχέση με την κοινωνία των πολιτών. Όταν μιλάμε για την κοινωνία των πολιτών, ορισμένες φορές μιλούμε για την οργανωμένη κοινωνία των πολιτών για επιχειρηματίες, συνδεκάτα κλπ. Την κοινωνία των πολιτών με την οποία μπορούμε να έχουμε ακριβώς ένα διάλογο λόγω της ενότητας εκπροσώπησής της. Αλλά υπάρχει μια πλατύτερη κοινωνία των πολιτών με την οποία θα πρέπει να αναπτύξουμε αυτή τη σχέση. Αλλά είναι σημαντικό η Επιτροπή των Περιφερειών καθώς και η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή να δραματίσουν ένα σημαντικό ρόλο ακριβώς σε σχέση με τους τοπικούς ε, φορείς από την άποψη του συντονισμού κάποιων εργασιών που ήδη έχουν υλοποιηθεί στον τομέα αυτό και που μπορούμε να θεωρήσουμε ενδιαφέρον στο πλαίσιο αυτού του διαφορεμένου διαλόγου. Θα ήθελα να ρωτήσω λοιπόν ποιο είναι ο ρόλο που έπαιξε η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή καθώ και η Επιτροπή Περιφερειών. Έχουμε ε, ήδη κάποιες, ε, ε, κάποια αποτελέσματα, κάποιες εμπειρίες στις οποίες να μπορούμε να αναφερθούμε έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Νομίζω ότι το θετικό αποτέλεσμα είναι αποτέλεσμα των κοινών προσπαθειών μας. Δεν είναι η Κομισιόν που θα πρέπει να συγχαρούμε, αλλά το σύνολο των εμπλεκομένων που κατέστησαν τη διαδικασία αυτή ε, επιτυχή. Για τον κύριο Ντέβα, να πω ότι προσπαθήσαμε εμείς να εμπλέξουμε το σύνολο των εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών. Σαν παράδειγμα, τα εμπορικά επιμελητήρια πήραν μέρος στο σύνολο της διαδικασίας αυτής. Επίσης και με τις οργανώσεις όπου αυτό ήταν εφικτό των ε, επιχειρηματιών. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο η Business Europe δεν μπόρεσε να πάρει μέρος, αλλά ελπίζουμε πάντα ότι κάποια στιγμή θα ενταχθούν στη διαδικασία. Προσπαθούμε όμως να εμπλέξουμε το σύνολο των συνιστοσών της κοινωνίας των πολιτών και όχι μόνο της ΜΚΟ ανάμεσα στους εταίρους που πήραν μέρος στο σύνολο της διαδικασίας έχουν εκπροσώπους και των συνεταιριστικών και ε, συνεργατικών οργανώσεων. Και όχι μόνο σε κοινωνικό επίπεδο αλλά και σε οικονομικό επίπεδο δραστηριοποιούνται αυτά. Έχουμε εκπροσώπους επίσης των πολιτικών Ινστιτούτων Ανάλογα με τις τοπικές πραγματικότητες έχουμε και άλλους παράγοντες οι οποίοι ε, εμπλέκονται και παίζουν ρόλο. Προσπαθήσαμε λοιπόν να κρατήσουμε το ευρύτερο δυνατό πεδίο σχετικά με τη συμμετοχή των ε, ε, εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών. Αυτό βέβαια δεν ανέβει τίποτα από τη σημασία της προσπάθειας που κάνουν οι ΜΚΟ, ιδιαίτερα και, και στον τομέα της δημιουργίας πλούτου. Για το μέλλον τώρα. Είναι σαφές ότι δεν μπορούμε εμείς να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία αυτή στη Βουδαπέστη και όλοι ευχαριστημένοι να γυρίσουν από εκεί που ξεκίνησαν. Νομίζω ότι ήδη έχουμε ξεκινήσει να αναπτύσσουμε μία σειρά προτάσεων, οι οποίες θα συζητηθούν με τον Επίτροπό μας την πρώτη εβδομάδα του Απριλίου, σχετικά με τη συνέχεια την οποία θα δώσουμε. Ήδη κατά τη διάρκεια των ομάδων εργασίας, της συνάντησης των ομάδων εργασίας την προηγούμενη εβδομάδα, ε, έγιναν, θα γίνουν μάλλον, θα, θα, θα προβλεφθούν δύο συναντήσεις με τους συναδέλφους που είναι υπεύθυνοι για τις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές. Θα δώσουμε στους συμμετέχοντες ε, τις ε, τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης για τις ε, δημοσιονομικές προοπτικές που είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε με τους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και όλους τους άλλους συμμετέχοντες σχετικά με τις τάσεις οι οποίες προδιαγράφονται έτσι ώστε οι απόψεις ε, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών να ληφθούν υπόψη. Δεν πρόκειται, θυμίζω, για μια διαδικασία διαπραγμάτευσης, αλλά για μια διαδικασία διαλόγου. Υπάρχουν χώροι, ιδιαίτερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για τις διαπραγματεύσεις αυτές, για τις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές. Δεν είναι αυτή η δουλειά μας. Θα υπάρξει επίσης και μια ειδική συνάντηση για την προετοιμασία για την τελική θέση δηλαδή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ελπίζω της Ευρωπαϊκής Ένωσης αργότερα και θα υπάρξει λοιπόν μια πρώτη δυνατότητα να ενημερώσουμε τους συναδέλφους οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για όλα αυτά και να τους μεταφέρουμε τα αποτελέσματα του διαφορετικού διαλόγου. Να θυμίσω επίσης ότι ο διαφορετικός διάλογος την επόμενη εβδομάδα θα διεξαχθεί ταυτόχρονα με το συνέδριο του, της συνάντησης ε, των τοπικών αρχών που γίνεται σε συνεργασία με την, Κοινωνική και Οικονομική, με την Περιφερειακή Επιτροπή και ένα ειδικό σεμινάριο το απόγευμα της 29ης θα ασχοληθεί ειδικά με τον ε, διαφορετικό διάλογο. Εδώ και δύο εβδομάδες συναντηθήκαμε επίσης και με τους συναδέλφους της Κοινωνικής και Οικονομικής Επιτροπής, οι οποίοι και αυτοί από την πλευρά τους προετοιμάζουν ένα ψήφισμα για το ρόλο της κοινωνίας των πολιτών. στα πλαίσια της συνεργασίας και των εξωτερικών σχέσεων γενικότερα. Αυτά είχα να πω και να πω επίσης ότι μετά τη Βουδαπέστη και στα πλαίσια των κεκτημένων της διαδικασίας θα ακολουθήσουν προτάσεις από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το τι θα ακολουθήσει. Ευχαριστώ Πρόεδρε, σας ευχαριστώ όλους για τη συμμετοχή σας και την εντατική μάλλον συμμετοχή. Διακόπτουμε λοιπόν τις εργασίες μας μέχρι τις 3 το απόγευμα στην ίδια αίθουσα.